Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Έχουμε αρκετούς συναδέλφους ώστε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Η ημερήσια διάταξη πρέπει να την έχετε. Υπάρχουν ε, αντιρρήσεις, ε, προβλήματα, παρατηρήσεις. Υπάρχουν δύο αλλαγές που θέλω εγώ να προτείνω. Για το σημείο 10 πρέπει να το αναβάλουμε γιατί ο κύριος Ιβαν δεν είναι στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα. Γίνονται οι προεδρικές εκλογές ε, την Κυριακή στην Ρουμανία, οπότε δεν μπορεί να είναι εδώ ο κύριος Ιβαν, οπότε θα το αναβάλουμε το 10 για τα κύρια, την έκθεση για, την, ε, για τα κύρια επιτεύγματα της στατικής ε, ΑΕ 2020, μετά το 11 του κυρίου Μπέλετ, που θέλει να μας μιλήσει για τη δικυβέρνηση του ίντερνετ, αλλά δεν μπορεί τη στιγμή που τον έχουμε βάλει, γιατί πρέπει να συναντήσει τον ε, βασιλιά του Βελγίου. Οπότε μας παρακάλεσε να αναβάλουμε το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης, οπότε θα το δούμε ως πρώτο αύριο το πρωί, πριν φύγει ο κύριος Μπέλετ και πάει στο βασιλιά. Έχει κανείς κάποιο πρόβλημα, όχι. Ωραία, εγκρίνεται λοιπόν η ημερήσια διάταξη με αυτές τις δύο αλλαγές. Πάμε στο σημείο 2, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης. Πρέπει να το έχετε λάβει. Μέχρι το τέλος της συνεδρίασης σήμερα. Σας παρακαλώ να μου πείτε εάν θέλετε κάτι να ζητήσετε για τα πρακτικά. Αν όχι, θα, θα θεωρηθούν ως εγκριθέντα. Πάμε στο σημείο 3 ανακοινώσει της Προέδρου ότι έχουμε web streaming στη σημερινή συνεδρίαση. Έχουμε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες, εκτός Μαλτέζικα, Σουηδικά, Λιθουανικά, Λετονικά και Εστονικά. Δεν έχουμε λοιπόν τις εστονικές γλώσσες, αλλά όλες τις υπόλοιπες ε, μπορείτε και να τις μιλάτε και να τις ακούτε. Ναι. Στις 5.30 έχουμε συνάντηση των συντονιστών. Το αποτέλεσμα θα το μάθετε σήμερα, θα σας στείλουμε email. Οπότε σήμερα το βράδυ ή το αργότερο αύριο το πρωί, πριν έρθετε στην, επόμενη, στην αυριανή συνεδρία, ελέγξτε τα email σας γιατί θα έχετε τα αποτελέσματα των συντονιστών. Οπότε, αύριο, ως πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, να μπορούμε να εγκρίνουμε και την απόφαση των συντονιστών. Υπάρχει μια μελέτη που έχουμε ζητήσει να γίνει για, ε, από τις υπηρεσίες έρευνας από την τελευταία θητεία, που ζητήθηκε από την τελευταία προηγούμενη θητεία, μια έκθεση για την α, ε, πολυπικιλότητα ε, στον τομέα της μουσικής. Ήταν στο παρελθόν μεγάλης σημασία σημασίας το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας. Η έρευνα τώρα ολοκληρώθηκε, η μελέτη ολοκληρώθηκε και θα παρουσιαστεί στην ομάδα νομικών υποθέσεων στις 3 την Δετάρτη το απόγευμα στις 2 του Δεκέμβρη. Αυτή η μελέτη λοιπόν, όποιος θέλει να την παρακολουθήσει, ε, στη Γιούρη την Τετάρτη στις 3. Ε, και τα λοιπά θα, υπάρχει και γραπτά, θα υπάρχουν και γραπτά αντίτυπα, θα τη λάβετε και από το, με email. Η διάσκεψη των Προέδρων έλαβε τρει τρεις αποφάσεις για τις ακροάσεις των επιτρόπων, αλλά υποθέτω ότι θα το έχετε ήδη ακούσει στις ομάδες σας. Οι ακροάσεις θα γίνουν από τις 11 μέχρι τις 15 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες και στις 18 και 19 Ιανουαρίου στο Στρασβούργο. Δύο ακροάσεις θα γίνονται παράλληλα, ταυτόχρονα, και κάθε ακρόαση τρει ώρε θα διαρκέσει. Στην αρχή είχαμε προβλέψει δυόμιση ώρε, αλλά επιμείναμε να είναι τρει, οπότε θα είναι τρει ώρες. ώρε. Και θα ε, μεταδίδονται και ζωντανά στο ίντερνετ. Έχουμε μια μήνυ ε, ολομέλεια την ε, Τρίτη στις 26 Ιανουαρίου και Εκεί το Κολέγιο των Επιτρόπων θα εγκριθεί ή όχι, αναλόγως, Έξτρα συνεδρίες, έξτρα ολομέλεια, συγγνώμη, στις 26 λοιπόν, επιπλέον. Και από την, ε, θα γίνει από κοινού με την ε, συνεδρίαση της ομάδας μας. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ε, τη Επιτροπή μα, συγγνώμη. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε, μπορείστε, μπορείτε όλοι να παρίσταστε. 26 λοιπόν Γενάρη, μείνει ε, ολομέλεια για τι ε, για να κλείσει και το θέμα αυτό. Ακόμη βέβαια εντάξει, ξέρουμε ποιος ε, θα είναι ο δικός μας ε, ε, ο Επίτροπος. Η Κύπρια Επίτροπος θα είναι αρμόδια για θέματα παιδείας, εκπαίδευσης, πολυγλωσσίας κτλ. Οπότε θα είναι και η βασική συνομιλητριά μας. Αλλά νομίζω ότι θα, έχουμε να, ασχοληθούμε και με την κυρία Κρός, γιατί θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της ε, ψηφιακής ατζέντα. Αυτοί οι δύο είναι, νομίζω. ΜΜΕ. Α, τα ΜΜΕ Εμεί τα έχουμε, εντάξει. Ωραία. Οπότε δύο τουλάχιστον ακροασει θα κάνουμε. Μία θα κάνουμε εμεί ε, δική μα για την εκπαίδευση, την, ε, τον πολιτισμό, τα ΜΜΕ και την πολυγλωσία και για τι υπόλοιπε, για την Έλλη θα συμμετάσχουμε. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Αύριο θα πάει μια μικρή αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας στη Στοκχόλμη. Θα προσπαθήσουμε το νωρίτερο λοιπόν να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση αύριο, έτσι ώστε όλοι να μπορείτε να διεκπαιρεώσετε τα εκκρεμή σα για να μην να σας πιάσει το σκοτάδι στη Στοκχόλμη, mm. ώσπου να φτάσετε. Πάμε στο σημείο 4 σε όλα τα στόματα βρίσκεται η Ευρωπαϊκή τώρα, χάρη στο Google. Ευτυχώς, εμείς εγκαίρως και χάρη στους Γάλλους συναδέλφους ε, ε, πιέσαμε ώστε να ξεκινήσει η Europeana, αυτή η online βιβλιοθήκη. Δεν θέλω εγώ να πω πολλά. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Τρίπελ που είναι και η συγγήτρια και θα την παρακαλέσω να μας κάνει έτσι μια πρώτη παρουσίαση για να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Παρακαλώ Χέλγκα. Αγαπητοί Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όντως υπάρχει μια αντιπαράθεση για τη ε, διευθέτηση, ε, το διακανονισμό του e-books από το Google και τώρα ήδη έχουμε περάσει ε, στη διευθέτηση του διακανονισμού και γι' αυτό έχει έρθει στο προσκήνιο η ε, βιβλιοθήκη μας η Ευρωπαϊκή και ελπίζω να έχει συνειδητοποιήσει και περισσότερος κόσμος στην Ευρώπη πόσο αποφασιστικό είναι για μας αυτό το σχέδιο για την Ένωση και για το μέλλον μας. Δεν νομίζω ε, ότι υπερβάλλω. Μιλάμε για μια Ευρώπη, πανευρωπαϊκή ε, βιβλιοθήκη που είναι το μεγαλύτερο και το πιο μεγαλεπίβολο σχέδιο στην ε, τομέα του πολιτισμού. Εκεί θα είναι η δραστηριότητά μας επίσης τα επόμενα χρόνια για να ε, καταφέρουμε να το κάνουμε το πιο φιλόδοξο πολιτιστικό σχέδιο. Όλα αυτά ξεκίνησαν όπως γνωρίζετε από το 2005 ως προσπάθεια υπήρξαν μερικές παιδικές ασθένειες από πλευράς τεχνολογίας και μέχρι να μπει το νερό στα βλάκι και μέχρι τώρα είναι 4,6 εκατομμύρια τα έργα που έχουν ψηφιοποιηθεί και μέχρι το 2010 θα είναι περίπου 10 εκατομμύρια. Είναι ψηφιακό σχέδιο, δεν πρόκειται μόνο για τα βιβλία, αλλά όλη η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης ε, χωράει εκεί. Είναι βίντεο, ταινίες, μουσική, ε, όλα αυτά που συνιστούν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά μπαίνουν στο διαδίκτυο και είναι στη διάθεση του κόσμου. Είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή από πλευρά ισότητα όλων των πολιτών που μπορούν να συμμετέχουν και από την άλλη έχει και πολύ μεγάλε απαιτήσει ποιοτικέ το σχέδιο αυτό. Δηλαδή να βλέπουμε το τι ε, συμπεριλαμβάνεται στη βιβλιοθήκη αυτό και όταν μπαίνει να είναι πραγματικά πολύ υψηλή ποιότητα. Για όλον τον κόσμο και για όλου του πολίτε παγκοσμίω, όχι μόνο στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά, είναι ανοιχτή για του πάντε. σε όλες τις επίσημες γλώσσες μας για τα 500 εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών. Λοιπόν, δεν, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένα μικρό σχέδιο, είναι πολύ φιλόδοξο πραγματικά και θα πρέπει να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια για να είναι καλή αυτή η προσπάθεια και να πετύχει. Μέχρι τώρα ε, τα έργα που είναι ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων, public domain το λένε στα αγγλικά αυτό, θα διατίθενται δωρεάν. Και διατίθεται σήμερα. Ωστόσο, υπάρχει εδώ ένα περίπλοκο σημείο, γιατί δεν έχουμε μόνο αυτά τα έργα, που να υπάρχουν ζητήματα ε, πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, αλλά αυτά είναι τα ορφανά, έργα, που δεν ξέρουμε πολύ καλά σε ποιον ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα. Εκεί πραγματικά χρειάζεται πολύ καλή και σε βάθος μελέτη, επαλήθευση και ένα μητρό όπου να συγκεντρώνονται όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι πολύ ε, ποιοτικό αυτό το ε, πρόγραμμα. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα Aero το οποίο συγκεντρώνει όλα αυτά τα έργα έτσι ώστε να ξέρουμε για με σαφείς κανόνες τι καθεστώς έχει κάθε φορά ένα έργο για να μην έχουμε παραβίαση του copyright και των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε αυτή την υπόθεση των e-books με την Google μπήκαν στο ψηφιακό σύστημα και κάποια βιβλία που ε, δεν ήταν ξεκάθαρο σε ποιον ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα, γι' αυτό και κατέληξαν οι περιπτώσεις αυτές στη δικαιοσύνη. Και περιμένουμε τώρα κρεμή ακόμα η δίκη. Ε, τώρα, η κατάσταση βέβαια στα ευρωπαϊκά κράτη δυστυχώς διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η Γαλλία έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο στη ψηφιοποίηση ε, και ε, στη διάθεση στην Ευρωπαϊκή πάνω από 40%. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία είναι περίπου στη μέση αλλά έχουμε και πολλά κράτη που δυσκολεύονται και αυτό έχει να κάνει και με την οικονομική τους κατάσταση. Και μέχρι τώρα δεν έχουν συνεισφέρει παρά σε πολύ μικρό βαθμό στην Ευρωπαϊκή και θέλουμε τα επόμενα έτη αυτό να αλλάξει για να υπάρξει μια πραγματική ψηφιακή βιβλιοθήκη πανευρωπαϊκή. Πολύ δε περισσότερο που είναι σημαντικό αυτό όχι μόνο για την κοινωνία της γνώσης και την κοινωνία της μάθησης στην Ευρώπη αλλά έχει επιπτώσεις και στην οικονομία, στην έρευνα, στον τουρισμό, στα μέσα ενημέρωσης. Όταν έχει κάνει ένα τέτοιο ψηφιακό πρόγραμμα ε, προσβάσιμο για όλους. Παναλαμβάνω, πρόσβαση για όλους τι σημαίνει αυτό, κατά τη δική μου άποψη τουλάχιστον, ότι αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται ε, παραβιάζοντας τα πνευματικά δικαιώματα και την προστασία τους, αλλά θα πρέπει να τα τηρούμε Και εντό παρεθέσεως πρέπει να σας πω ότι του χρόνου θα μας απασχολήσει πάρα πολύ αυτό το θέμα και μεταξύ διαφόρων επιτροπών του Κοινοβουλίου. Τώρα, α πούμε, η κυρία Ρέντεν κατέθεσε μια ανακοίνωση όπου ζητάει ρητά εναρμόνιση, παρακαλώ, ε, το ευρωπαϊκού δικαίου για τα πνευματικά δικαιώματα. Αυτό είναι πάρα πολύ επίμαχο ε, μεταξύ των ενδιαφερομένων και η δική μας Επιτροπή που ενέχεται εκεί και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και Εσωτερικής Αγοράς και η Βιομηχανία. Όλες αυτές οι επιτροπές ασχοληθούν με το θέμα του χρόνου και θα είναι έτσι πάρα πολύ καυτό και ακαθόδες να δούμε πώς θα το ρυθμίσουμε σωστά. Από την άλλη, βεβαίως, είναι σαφές, θέλουμε κάποια έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα να μπουν και αυτά στη βιβλιοθήκη για να μην έχουμε μια μαύρη τρύπα για ολόκληρο τον 20ο και 21ο αιώνα. Απλώς θα πρέπει να δούμε πώς ε, ε, θα ε, πληρώνει κανείς για να έχει πρόσβαση σε αυτά τα έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Να συνοψίσω λίγο. Κατά την άποψή μου, όλα αυτά συνηγορούν υπέρ της εύκολης, απλής προσβάσεως και προς το να είναι ένα μεγάλο εγχείρημα και φιλόδοξο πολιτισμικό ε, από τη μια, από την άλλη όμως να μην παραβιάζουμε την κείμενη νομοθεσία και αν καταλήξουμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε τη νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα θα πρέπει να υπάρχουν πολύ καλοί κανόνες και πολύ σωστοί γιατί θεωρώ εγώ καταρχήν ότι ε, για να λειτουργεί καλά μια δημοκρατική κοινωνία και μοιραία και στο ίντερνετ, γιατί δεν μπορεί να είναι διαφορετικό το διαδίκτυο από τον πραγματικό κόσμο, χρειάζονται κανόνες και για τα πολιτιστικά θέματα και βέβαια δεν θέλω το διαδίκτυο να κλείσει, ναι, να υπάρχει μια πολιτική διήθηση, δεν είμαστε εδώ ούτε Κίνα ούτε Ιράν, αλλά να υπάρχουν καλοί κανόνες, να σταθμίζουμε τα πράγματα, τα έργα των ε, δημιουργών, των ε, ε, καλλιτεχνών που και εκείνοι θα πρέπει να πληρώνονται για το έργο τους ακόμα και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Όλα αυτά είναι ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Κάτι άλλο που με χαροποιεί και θα το βρείτε και στην έκθεσή μου και θα πρέπει να το συνεχίσουμε, είναι ότι πέρσι και τα τελευταία χρόνια είχαμε μια ομάδα πολύ ψηλού επίπεδου εμπειρογνωμόνων από διάφορες ψηφιακές βιβλιοθήκες της Ευρώπης που ε, ασχολήθηκαν διαμακρό με το θέμα αυτό και θα πρέπει να ανανεωθεί η θητεία της ομάδας γιατί είναι πολύ Πολύτιμέ οι συμβουλέ τους και πολύ ψηλού επίπεδου για όλα αυτά τα θέματα που είναι και περίπλοκα και πώς μπορούμε να βρούμε ένα καλό ευρωπαϊκό δρόμο για να αντιμετωπίσουμε αυτή την ιστορία. Τώρα, για να έρθω στην πολιτική συζήτηση, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση και οι άτομα με αναπηρίες, θα τα συζητήσουμε αυτά αργότερα στη συνέχεια. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την προστασία των ε, πνευματικών δικαιωμάτων, ε, διάφορα μέτρα συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων αυτών, ποια είναι τα υπέρ, ποια είναι τα κατά, να έχουμε ένα σαφή ορισμό για τα λεγόμενα ορφανά έργα, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε πώ ορίζεται αυτό. Σα είπα προηγουμένω πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια σαφή βάση δεδομένου και γιατί χρειάζεται ε, οπωσδήποτε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, πρόγραμμα αν θέλετε τώρα να περάσουμε στα διοικητικά και τα διαδικαστικά, την τελευταία φορά που συζητήσαμε τη βιβλιοθήκη αυτή, ήρθε και το μεγάλο ζήτημα της χρηματοδότησης και είναι σαφές ότι τα πολιτιστικά ιδρύματα στα διάφορα κράτη-μέλη θα πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη και από τον ίδιο προϋπολογισμό τους να συνεισφέρουν, αλλά βεβαίως και οι κρατικοί εκάστοτε προϋπολογισμοί, ο καθώς επίσης και ο ευρωπαϊκός προπολογισμό. Μέχρι τώρα έχουμε το πρόγραμμα, το e-content ε, plus, που χρηματοδότησε την προσπάθεια αυτή και θα συνεχιστεί στο μέλλον, αλλά αν δούμε την περίοδο μετά το 2013, θεωρώ και θα το συζητήσουμε ότι θα ήταν επιθυμητό από τη νέα στρατηγική της Λισαβόνας για το πώς θα κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ανταγωνιστική ε, οικονομική δύναμη και σύγχρονη, τότε θα πρέπει ένα τμήμα του προπολογισμού της Στρατηγικής Λισαβόνας να πάει ε, στην ψηφιοποίηση του κοινοτικού κεκτημένου στο τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Γιατί είναι πραγματικά κοινή μας κληρονομιά. Επίσης, σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα, γιατί όχι. Βεβαίως πάντα με καλές ε, ε, προϋποθέσεις, με καλές διαπραγματεύσεις και καλό αποτέλεσμα, αλλά να το προωθήσουμε αυτό, να κάνουμε μια ενημερωτική εκστρατεία. Join Europeana. Και όχι μόνο από κρατικού πόρους, γιατί σας είπα ότι βεβαίως θα πρέπει να γίνει αυτό και σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά καλό θα ήταν και πάνε στα πάρα πολύ ωραίο να έχουμε και ιδιωτικά κονδύλια, μεγάλα ιδρύματα, Ινστιτούτα, γιατί όχι και μεγάλες επιχειρήσεις. Ε, θα μπορούσαν να συμμετέχουν, γιατί μετά κάνουν και διαφήμιση ε, στο Google και αλλού. Δεν θα πρέπει η Ευρώπη εδώ να χάσει το τρένο της τεχνολογίας, να κάνουμε κάτι καλό, να συνεργαστούμε δημόσιος και ιδιωτικός τομέας υπεύθυνα και σωστά. Λοιπόν, επιθυμώ να γίνει μεγάλη συζήτηση για αυτό το μεγάλο σχέδιο, για να λυθούν και τα ανοιχτά ζητήματα και οι λεπτομέρειες, αλλά να δημιουργηθεί και έτσι μια ορμή πολιτική, γιατί υπάρχει και η ε, ιστορία του ανταγωνισμού με τη Google πώς μπορούμε να στήσουμε σωστά αυτό το πρόγραμμα, να βρούμε τα απαραίτητα κονδύλια και να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών πολιτιστικών φορέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτη-μέλη και Ευρώπη. Και έτσι ελπίζω τα επόμενα έτη βιβλιοθήκη αυτή να γίνει μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή η ιστορία για την Ευρωπαϊκή είναι πάρα πολύ επίκαιρη. βλέπουμε τα σχέδια του Google καθημερινά. Έχει βρει τώρα μια λύση που δεν μπορώ να πω ότι μας ικανοποιεί και σε αυτό το σχέδιό μας για τη Ευρωπαϊκή θα πρέπει να είμαστε πραγματικά παράδειγμα και να δίνουμε το καλό παράδειγμα, να δούμε τι ζητάμε και από τους άλλους. Τα περίφημα ορφανά έργα όπως τα χαρακτήρισες θα πρέπει να τα δούμε και να δείξουμε στην Google πώς το κάνουμε. Ε, εκείνοι έχουν την αμερικανική νοοτροπία ε, που ε, είναι κτήρα μέτρο αντίθετα με τη δική μας. Και εμεί θα πρέπει να, σεβόμαστε και να διασφαλίζουμε πάντα την πνευματική ιδιοκτησία, τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Είναι μεγάλο μας μέλημα. Βεβαίως να είναι όσο γίνεται ανοιχτή και δωρεάν η πρόσβαση, χωρίς όμως αυτό να είναι των δικαιωμάτων των δημιουργών. Εύκολο δεν είναι, αλλά είναι πολύ ο κόσμος που ασχολείται με αυτή την νομοθετική προσπάθεια και ελπίζω να ευοδοθεί. Να δώσω αμέσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή πρώτα στους συναδέλφους. Ε, όχι, τους συναδέλφους πρώτα. Ναι, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Χέλγα Τρίπελ για το σχέδιο της έκθεσης, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό, περιλαμβάνει πάρα πολλές πτυχές που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή. Καλύπτονται λοιπόν όλα αυτά με πολύ σωστό τρόπο. Όντως, καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή να αποτελέσει αυτό το μεγάλο πολιτικό, πολιτισμικό ε, project της Ευρώπης. Σε σημαντική προπόθεση βέβαια είναι να μην ε, το προωθήσουμε μόνο το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν και να είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό, αλλά και τα κράτη-μέλη να εμπλακούν σε όλη αυτή τη διαδικασία και να είναι υπεύθυνοι, γιατί θεωρώ ότι και τα 27 κράτη-μέλη θα πρέπει να δώσουν την δέσμευσή τους ως προς την Ευρωπαϊκή ε, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία. Ήδη συμβαίνει αυτό, γιατί το, ε, το, αν συμβάλλουν όλοι μπορούν, θα μπορέσει το project αυτό να είναι επιτυχές για να μπορέσει να αποτελέσει και μια ανταγωνιστική λύση για το Google Books κτλ. Και πιστεύω ότι ίσως στο σχέδιο έκθεσης ή στη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας θα έπρεπε να καταστήσουμε σαφές ότι η ευθύνη των κρατών μελών ε, υπάρχει, υφίσταται και υπάρχει και μια κοινή πολιτική, ε, κοινοτική ε, για να προωθηθεί η πολιτιστική κληρονομιά και να είναι προσβάσιμη σε όλους την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η προσβασιμότητα, κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι Όπω και για τι ανοιχτέ βιβλιοθήκε, τι κλασικέ δηλαδή βιβλιοθήκε, όπου πάει κανεί, μπαίνει μέσα και ε, δανείζεται τα βιβλία ή τα CD ή ε, μια ταινία. Η ευθύνη λοιπόν για, για την βιβλιοθήκη αυτή θα πρέπει να είναι, ε, να είναι προσβάσιμη, όπως είναι και στις υπόλοιπες βιβλιοθήκες. Αυτό είναι σημαντικό θέμα. Είναι σημαντική οικονομική πρόκληση, χρηματοδοτική, αλλά αν όντω θέλουμε να χωρίσουμε τη θέση μα από το Google και θέλουμε να αποφύγουμε την κλασική ας πούμε διαφήμιση, αν θέλουμε να αποφύγουμε λοιπόν αυτό, και για να διαχωρίσουμε τη θέση μας από το Google και ως προς αυτό θα πρέπει να είναι όσο δυνατόν πιο μικρή η οικονομική συμβολή αν όχι δωρεάν η ε, πρόσβαση. Υπάρχει βέβαια και το θέμα της ε, ποιότητας ε, και εκεί θα πρέπει να δείξουμε ποια είναι ε, η δική μας θέση. Γιατί αν εμείς τώρα έπρεπε να πάρουμε λεφτά για την Ευρωπαϊκή, τότε όντω το Google Books θα ήταν φυσικά πιο, η πιο εύκολη λύση, η πιο α, χρήσιμη. Και αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σίγουροι ότι και η Ευρωπαϊκή θα είναι σαφώς ποιοτική και πιο ποιοτική ακόμη από τα Google Books και για την κατηγοριοποίηση των έργων και των βιβλίων ε, ε, στο Google πραγματικά έγιναν τεράστια ε, λάθη. Υποθέτω ότι δεν θα γίνουν αυτά στην Ευρωπαϊκή και ακριβώς θα διασφαλιστεί η ποιότητα ως προς αυτό για να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε τη δική μας θέση από αυτούς. Και επίσης να πω ότι είναι πολύ σημαντικό που αναφέρετε στην έκθεσή σας το θέμα των συμπράξεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενώσουμε επιχειρήσεις, ιδρύματα, να εμπλακούν και οικονομικά στην όλη αυτή η διαδικασία. Αλλά θα πρέπει να πούμε σαφώς άλλη μια φορά ότι αυτή η κλασική χρηματοδότηση μέσω διαφημίσεων όπως γίνεται μέσω άλλων ε, ίντερνετ ε, δεν θα πρέπει να ισχύει για την Ευρωπαϊκή. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το πούμε σαφώς, να δώσουμε το μήνυμα ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός ως προς, αυτό, ως προς αυτό για την Ευρωπαϊκή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καβαντά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την εισηγήτριά μας την κυρία Όλγα Τρούιπελ γιατί ναι, ε, ε, πραγματικά έχει πει πάρα πολύ σωστά πράγματα στην έκθεση αυτή που αποτελούν μια ορθή βάση εργασίας, πράγμα όχι και τόσο προφανές ε, και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να εκφράσω την μεγάλη ικανοποίηση που αισθάνθηκα διαβάζοντας την βάση της εργασίας σας. Αλλά βέβαια οι δυσκολίες τώρα αρχίζουν για όλους εμάς. Κυρία Πρόεδρε, κατά αυτή την έννοια θα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι εδώ Ε, σε αυτή την Επιτροπή που δεν διαθέτει τα ίδια μέσα ε, και να πω από τι άλλες Επιτροπές του Ιδίου Κοινοβουλίου και να πω ότι αυτό ε, αποτελεί ήδη ένα αρνητικό σημείο Πρόκειται λοιπόν για ένα μήνυμα ε, προκατάληψης ε, το οποίο θα πρέπει να διορθώσουμε. Δηλαδή η Ευρώπη θέλει βεβαίως και κανόνες θεσμοθετημένους αλλά θέλει και ψυχή, θέλει και πνεύμα. Γι' αυτό λοιπόν δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο στην έκφραση των πολιτισμών και τονίζω γενική πληθυντικού των πολιτισμών της Υπήρου. Το δεύτερο, η δεύτερη παρατηρήσή μου αφορά άμεσα την έκθεσή σας, κυρία ε, Τρύπελα. Από τη σύνθεση κατανοούμε κάτι, μια ιδέα υποβόσκουσα, αλλά πολύ σημαντική. Δηλαδή, τα μέσα δεν είναι ουδέτερα ε, και ε, ειδικά τα πιο μοντέρνα στοιχεία δεν είναι απαραίτητα σύμμαχοί μας. Θέλω να πω με αυτό ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε όλοι μια οικονομική βάση έτσι ώστε να επιβιώσουμε. Και πέρα από το δημόσιο τομέα υπάρχει και ο ιδιωτικός τομέας και δημιουργείται λοιπόν σε όλες τις χώρες και στη δικιά σας περιοχή και στη δικιά μου και παντού μία αγορά πολιτισμού η οποία επιτρέπει την αγορά και την διάδοση των έργων τέχνης. Επομένως, αυτή είναι μια πολύ ε, σημαντική ιδέα που πρέπει να φαίνεται και στην έκθεσή σας, δηλαδή ότι χρειάζεται και η τέχνη και ο πολιτισμός οικονομική βάση ε, και βεβαίως προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Και επίσης, τι θέλουμε να κάνουμε τώρα. Θέλουμε να μεταφέρουμε σε άλλη βάση όλα τα γραπτά στοιχεία, τα ηχητικά ε, στοιχεία και τα οπτικοακουστικά γενικά ε, σε υπόβαθρα, ε, σε τρόπους ε, υποστήριξης που θα είναι πολύ πιο εύκολα αναγνώσιμα στο μέλλον. Δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι ο πολιτισμός ποτέ δεν πρόκειται να δώσει τη θέση του, τη σημαντική του θέση προς οποιοδήποτε τρόπο στήριξης. Είναι μια αγγλοσαξονική ιδέα που λέει ότι τα μηχανήματα μπορεί να είναι πιο σημαντικά από την τέχνη ή από το περιεχόμενο που μεταφέρουν. Όχι. Η τέχνη, ο πολιτισμός είναι πάντα πάρα πολύ σημαντικός και θα κρατήσει την ψυχή του όπου κι αν είναι καταγεγραμμένος. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε αυτό να το υπογραμμίσουμε. Επίσης οι δημιουργοί είναι αυτοί οι οποίοι οργανώνουν την αγορά και ε, την αγορά του πολιτισμού και άρα πρέπει να τους στηρίξουμε με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων κλπ. Επίσης, θα πρέπει να προστατεύσουμε τα έργα τα οποία έχουν μεταφερθεί σε άλλη μορφή, να τα προστατεύσουμε, λέω, από οποιαδήποτε, ε, οποιαδήποτε φθορά. Εγώ προσωπικά έζησα ε, σαν πολύ νέος ε, δημοσιογράφος την εποχή που μας έλεγαν ότι ε, το μαγνητοσκοπημένο υλικό πάνω σε κασέτα, σε βιντεοκασέτα δεν θα πάθαινε ποτέ τίποτα. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά που είχαμε καταγράψει σε κασέτες βίντεο αυτή τη στιγμή μερικές φορές δεν διαβάζονται καν και δεν είμαι πια και μαθουσάλας. Τώρα, η δουλειά μας εδώ, ε, η δουλειά των Ευρωπαίων, είναι να μην αφήσουμε τον πολιτισμό σε ένα μονοπόλιο, ιδιαιτέρως δε ιδιωτικό μονοπόλιο, να το κρατήσει λοιπόν και όπως θέλει εκείνος ο τομέας να το μεταφέρει και να, σε ψηφιακή βάση να το ψηφιοποιήσει. Δηλαδή εμείς πρέπει να δώσουμε μια ικανοποιητική λύση απέναντι, εναλλακτική λύση απέναντι στην Αμερικάνικη φύρμα που έχουμε επανειλημμένα αναφέρει εδώ. Και βλέποντας πάντα ε, προς την πλευρά του Google, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρχει λογοκρισία, δεν θα υπάρχουν λάθη, όπως είπε προηγουμένως η συνάδελφος, γιατί είναι πολύ σημαντικά, και ούτε μερική μεταγραφή. Προ υποσημείωση επίσης, αλλά φαντάζομαι ότι συμφωνούμε όλοι, να πω ότι η βάση μεταβίβασης θα πρέπει ε, να συμφωνηθεί και από του ε, ε, και από τους κανόνες που καλύπτουν τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Πιστεύω ότι στο σύνολο του θέματος αυτού, κυρία Πρόεδρε και κυρία Εισηγήτρια, πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα το Αεροπεάνα είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα, αλλά ξεκινάει 10 χρόνια αργότερα από ό,τι θα έπρεπε. Γιατί ήδη έχουν πάρει σημαντικό προβάδισμα ε, οι Αμερικανοί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο τρόπος ανάγνωσης ε, είναι διαφορετικός πλέον. Ε, είναι ε, μέσα από αυτήν την Αμερικάνικη φίρμα και το βλέπουμε και στο e-book και σε άλλες προσπάθειες. Είναι μερική, είναι μεροληπτική πολλές φορές, άρα και επικίνδυνη. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το εμποδίσουμε αυτό, δεν ξέρω ποιο είναι το νομικό εργαλείο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τώρα ή στην επόμενη φάση. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ομάδα η οποία θα σας βοηθήσει έτσι ώστε να προχωρήσουμε στο μέλλον προσεκτικά. Και κατά αυτή την έννοια ναι, θα υποβάλω με κάποιες τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Καβαντά. Κύριος Μάρτιν. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Συναρπαστικό το θέμα. Μετά το βραβείο Λουξ, που δυστυχώς δεν μπόρεσα να βοηθήσω όσο θα ήθελα γιατί με ταλαιπωρεί μια ασθένεια. Είναι μια τεράστια υπόθεση η Ροπεράνα. Η κυρία Τρούπελ, ε, στα χέρια της κυρίας Τρούπελ είναι σε εξαίρετα χέρια και η πρόεδρος μας και πολλοί από εμά ε, συμμετέχουμε από καρδιάς. Τα θέματα των ε, πνευματικών δικαιωμάτων σίγουρα θα τα κάνετε σωστά. Τώρα για τη διαφήμιση στο διαδίκτυο είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και εγώ θα επικεντρωθώ σε δύο θέματα που αναφέρονται και στη συζήτηση, στην έκθεσή σας, ε, παράγραφο 19, 20 και 21 του σχεδίου έκθεσης. Σε αυτό το σχέδιο ε, Ευρωπαίανα είναι μία από τις ευκαιρίες ε, να έχουμε πάρα πολύ θετικό αποτέλεσμα υπέρ του ευρωπαϊκού ιδεώδους από πού ερχόμαστε, πού πηγαίνουμε, τι μας ενώνει, τι μας χαρακτηρίζει και να το προβάλλουμε αυτό. Και σας παρακαλώ, σας παρακαλώ όμως στη διαδικασία να γίνει πιο διαφανής η διοίκηση και η χρηματοδότηση από ό,τι μέχρι σήμερα. Εγώ δεν θα ήθελα απλώ πολύ περισσότερα χρήματα, πάρα πολύ περισσότερα χρήματα, αλλά να είναι και υποδειγματικό για το πώς θα διαχειρίζεται κανείς αυτά τα κονδύλια. Θα το θεωρούσα τραγικό να κατακαιρματιστεί στον προπολογισμό. Κυρία Τρούπελ, έχετε πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από μένα, αλλά λίγη έχω μαζέψει και εγώ στην Επιτροπή Προπολογισμού. Τα παίρνουμε από εδώ και από εκεί, ε, είναι τελείω ε, αδιαφανής η διαδικασία, τα ρίχνουμε στο ίδιο καζάνι και ορισμένοι που τους απορρίπτω και εγώ στις απόψεις τους ε, θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν, να το ιδιοποιηθούν αυτό ως προπαγάνδα. Θα μπορούσαμε λοιπόν λίγο πιο συγκεκριμένα ε, να το γράψουμε στην έκθεσή σας και θα κάνω και τροπολογίες. Και θα το φέρω και εγώ ως γενικό αίτημα. Υποδειγματικό όχι μόνο στην ουσία αλλά και στον τύπο, να φαίνεται και τίμιο, δηλαδή όχι μόνο να είναι besprochen haben. Ε, δεύτερο σημείο, η διαφήμιση προς τα έξω. Ε, δεν ε, έχουμε κανένα όφελος αν φτιάξουμε ένα καταπληκτικό σχέδιο και δεν το μάθει ψυχή. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα, είναι πάρα πολύ πολύτιμα όλα αυτά που προτείνουμε. Έχει μεγαλώσει περισσότερο από ό,τι περιμέναμε και αυτά τα 10 εκατομμύρια ε, ε, βιβλία και κείμενα μέχρι το μέσο του επόμενου έτους. Ωραία. Θα ήθελα όμως και πολλοί πολίτες της Ένωσης, άνδρες και γυναίκες, να το μάθουν ότι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα. Και εδώ υπάρχει αυτό το θέμα της ΔΕΙΤ, ε, σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και είναι πολύ επίμαχο. Ένα καλό της οικονομικής κρίσης είναι ότι περσεύει χώρος για διαφήμιση. Αν θεωρήσουμε ότι η ζωή είναι ποδόσφαιρο και όλα τα υπόλοιπα είναι ε, απλώς οδοντόκρεμες, ε, κοιτάξτε, του χρόνου έχουμε ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχαμε τρομερούς αγώνες. Arsenal, Chelsea και Βαρκελόνη, Μπάρτσα, Ρεάλ Μαδρίτης. Είχαν από πίσω τους ε, διαφημιστικά πανό και μάλιστα πολλά άδεια. Δεν μπορούμε εμείς να το βάλουμε αυτό το πρόγραμμα Europeana, εκεί διαφήμιση, με πολλαπλασιαστές όπως ονομάζονται του μηνύματος, με διαφημιστές, να μας βάλουν τη διαφήμιση μας εκεί δωρεάν. Ε, γιατί στη Βαρκελόνη ε, έγραφε UNICEF από πίσω. Ή στις φανέλες τους ας πούμε, δεν μπορεί να γράφει Europeana. Γιατί όχι. Είναι πολύ καλό το πρόγραμμα, να είναι καλή η διοίκηση και η διαχείριση και όσο μπορώ να σας βοηθήσω κι εγώ. Ευχαριστώ. Ναι, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συγχαρώ την κυρία Τρούπελ για την έκθεσή της η λεπτομερής αυτή έκθεση είναι μια έκθεση στην οποία, με την οποία συμφωνήσαμε. Είδαμε πόσο μεγάλο εύρος έχει το πρόγραμμα αυτό και πόσο περήφανοι θα μπορέσουμε να είμαστε. Νομίζω ότι είναι δικό μας παιδί, της δικής μας επιτροπής. Και είμαι σίγουρος ότι η κυρία τρύπελ θα, με την κυρία Τρούπελ βρίσκεται στα καλύτερα χέρια ε, το πρόγραμμα αυτό. Για τη χρηματοδότηση είχα κάποια ερωτήματα. Βλέπουμε ότι το project αυτό πραγματικά είναι πολύ ευρύ και προφανώς θα χρειαστεί και μεγάλα κονδύλια. Η συγγήτρια μας μίλησε για τις, ε, για συμπράξεις, για τους σπόνσορες, για τη συμπερίληψη των κρατών μελών στην όλη αυτή διαδικασία. Οπότε πρέπει να υπάρξει και ε, κατανομή οικονομικών βαρών προφανώς. Ε, αυτό θα ήταν καλό και προς όφελος του στόχου μας. Και θα ήθελα να θέσω το ερώτημα, αν στον προϋπολογισμό για το από 2007 μέχρι 2013 πόσο υψηλό είναι το ποσό το οποίο θα αποδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προβλέπεται για το φανταστικό αυτό project, το οποίο δεν αφορά μόνο την ε, προστασία της ε, πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά διατήρηση και της ευρωπαϊκής ε, ταυτότητας. Ευχαριστώ. Ich möchte mich zunächst einmal dem Dank meiner Να ευχαριστήσω για την έκθεση. Η κυρία Τρούπελ νομίζω ότι έχει κάνει πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Μια άποψή μου, μια σκέψη μου να πω. Την είπατε και εσείς βέβαια κυρία Τρούπελ. Ο κανόνας, ποιοι κανόνες θα ισχύσουν για την Ευρωπαϊκή. Είναι σημαντικό αυτό γιατί πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε στο ίντερνετ με το copyright, με τα δικαιώματα τα πνευματικής ιδιοκτησίας. Έχουμε τον πραγματικό κόσμο, έχουμε και τον ψηφιακό κόσμο πρέπει να πείσουμε τους νέους να χρησιμοποιούν τον κόσμο του ίντερνετ με, σωστό τρόπο. Να μην αποφύγουν δηλαδή να πηγαίνουν σε μια κανονική βιβλιοθήκη και να παίρνουν ένα βιβλίο να δανείζονται. Υπάρχουν και εκεί κανόνες. και νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξουμε ώστε η Ευρωπαϊκή να τύχει διαχείρισης σωστή Ελεύθερη φυσικά πρόσβαση, ε, το κατά πόσο θα είναι δωρεάν ή όχι είναι άλλο ένα θέμα η χρηματοδότηση ενός τέτοιου project επίσης είναι σημαντικό, αν δηλαδή θέλουμε να προωθήσουμε τη δημιουργικότητα, να διασφαλίσουμε τα πνευματικά δικαιώματα, το είπε και ο κύριος Καβαντά πολύ σωστά για τη νέα δημιουργικότητα που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει, δεν υπάρχει στον πραγματικό κόσμο, υπάρχει στον ψηφιακό κόσμο και από κάπου πρέπει να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι που δημιουργούν συνέχεια. Αυτό σημαίνει κόστος. Οπότε πρέπει να έχουμε σημαντικό, σημαντικούς και αυστηρούς κανόνες για το τι θα γίνει με το copyright και πώς θα χρηματοδοτηθεί όλο αυτό. Και αυτό βέβαια πρέπει να το δούμε παράλληλα με τα ουσιώδη. Θα είναι νομίζω ένα πολύ καλό επιχείρημα. Και θα πρέπει να ασχοληθούμε εντατικά τον επόμενο καιρό με αυτό, γιατί το πρόγραμμα αυτό πραγματικά αξίζει τον κόπο. Και ίσως θα πρέπει να δώσουμε πολύ περισσότερα από ό,τι τώρα σκεφτόμαστε. Ευχαριστώ. Pääsee, pääsee kärryille. Eli tämä on Ευχαριστώ πολύ. Ε, πρόκειται για μια πάρα πολύ καλά δομημένη έκθεση για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Τα προβλήματα όμως ε, εδώ ε, έχουν διαφορετικές διαστάσεις στο καθένα. Όπως άλλωστε ανέφερε και η συγκήτρια, η Γερμανία, οι κατοχώρες, η Γαλλία, ή το Ηνωμένο Βασίλειο κάνουν πολλά, αλλά όταν έρχεται κανείς από μία μικρή χώρα και όπου μιλιέται μια μικρή γλώσσα είναι λίγο δύσκολο να έχει πρόσβαση στα κονδύλια και επομένως ε, στην προκείμενη περίπτωση θα βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση για τις μικρές χώρες όσον αφορά την εναρμόνιση των πνευματικών δικαιωμάτων του copyright. Η νέα γενιά τα βλέπει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Θεωρεί ότι έχει δικαιώματα ε, στο ίντερνετ και ότι τα δικαιώματά της δεν έχουν όρια. Όμως πιστεύω ότι πολλοί μεταξύ ημών πιστεύουν, θεωρούμε ότι ο δημιουργός πρέπει να πληρωθεί με κάποιο τρόπο, γιατί ο, δημιουργός θέλει να ζει από, από το πνευματικό του έργο, την πραγματική του δημιουργία και όχι από οποιασδήποτε επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις. Και Επομένως, ε, οι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν θέλουν οπωσδήποτε να αμείβονται για τη δημιουργία τους. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που πιστεύουν ότι αφού πέσαμε πάνω στο έργο ας το ακούσουμε, ας το διαβάσουμε και από εκεί και πέρα αργότερα ίσως σκεφτούν λίγο και την ε, οικονομική διάσταση του θέματος. Και βεβαίω ε, καταλαβαίνετε ότι όπω ε, και ο κάθε επιχειρηματία ξεκινάει με μια μικρή επιχείρηση και σιγά σιγά μεγαλώνει, έτσι και ο δημιουργό θα ξεκινήσει με μια μικρή α το πούμε ε, επιχείρηση και θα μεγαλώσει. Απ' την άλλη πλευρά μην ξεχνάτε ότι διανύουμε εποχή οικονομική κρίση και οικονομική ύφεση και από τη στιγμή που οι δημιουργοί δεν βρίσκουν πλέον χορηγού, δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στο χρήμα, τότε θα πρέπει το δημόσιο ή θα πρέπει ο κόσμο να πληρώσει πληρώσει. Ε, βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις ε, όπου μπορεί κανείς ε, να ακούσει, να διαβάσει τα έργα δωρεάν όπως είναι οι βιβλιοθήκες, αλλά αυτό είναι μια διαφορετική περίπτωση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρώπη ε, βασίζεται στην αρχή της πολυγλωσσίας και στην αρχή της διαφορετικότητας και η διαφορετικότητα αυτή θα πρέπει να βρει τρόπους να εκφραστεί. Κατά αυτή την έννοια συμφωνούμε απολύτως με την έκθεση. Αλλά το οικονομικό ζήτημα και το ζήτημα του copyright είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ και δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να το λύσουμε. Στις σκανδιναβικές χώρες από που προέρχομαι έχουμε ακόμα και πολιτικά κόμματα τα οποία είναι υπέρ της πειρατείας και κατά ε, του copyright και επομένως πρέπει να βρούμε τρόπους να στηρίξουμε τους καλλιτέχνε, όπως και εγώ θέλω να τους στηρίξω προσωπικά. Αγαπητέ συνάδελφοι, είπατε ότι δεν είστε ε, οπαδός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είστε, γιατί αλλιώ πού θα ήταν η επικοινομορφία και η διατήρησή της. Κυρία Βερία. Euh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την κυρία Τρούιπελ γιατί πιστεύω ότι θέτει ορθώς τα κυριότερα θέματα η έκθεση αυτή. Ορισμένες παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Πιστεύω στο ευρωπαϊκό μοντέλο. Πιστεύω ότι υπάρχει και κοινωνικό μοντέλο αλλά και πολιτιστικό ευρωπαϊκό μοντέλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πιστεύω ότι υπάρχει μια ε, ευρωπαϊκή ταυτότητα, όπως άλλωστε δεν θέλω και την, ε, να δεχτώ και την έννοια της εθνικής ε, ταυτότητας. Ο πολιτισμός, όπως έλεγε ο κ. Καβαντά προηγουμένως, έχει ψυχή, κινείται, προχωράει. Επομένως, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι ένας πολιτισμός ο οποίος δέχτηκε νέα στοιχεία που τον εμπλούτησαν στη, διάρκεια της ιστορίας του. Νομίζω ότι με, το, με την Ευρωπαϊάνα εκφράζουμε πραγματικά δίνουμε μάλλον μια ορθή απάντηση σε όλα τα διακυβεύματα τα οποία κρύβονται πίσω από το θέμα της, ε, ε, ε, του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ε, υπόθηκε προηγουμένως ότι ο πολιτισμός δεν είναι στις ευρωπαϊκές αρμοδιότητες ε, και εγώ λέω ευτυχώς γιατί όσο το θέμα του ανταγωνισμού θα είναι βάση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος τότε ε, τα οικονομικά θα είναι αυτά τα οποία θα βρίσκονται στο κέντρο αυτού του ευρωπαϊκού οικοδομήματος ε, και δεν είναι τέτοιο διακύβευμα ο πολιτισμός. Γι' αυτό λοιπόν δεν αλλάζω και εγώ γνώμη για τη συνθήκη της Λισαβόνας, αυτήν που είχα εξακολουθώ να την έχω. Πάντως αυτό που έλεγε ο κύριος Καβαντά είναι αλήθεια, δηλαδή ότι υπάρχουν και οικονομικά στοιχεία γύρω από την πνευματική δημιουργία. Όμως δεν θα πρέπει να συρρυκνώσω με τον πολιτισμό και την πολιτιστική παραγωγή και δημιουργία ε, σε θέματα ε, οικονομικά και σε θέματα αγοράς τούτων λεχθέντων πιστεύω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο τι είναι και η οικονομία. Η οικονομία δεν είναι απαραίτητα εμπορεύσιμη. Ε, και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό στον πολιτισμό. Ε, του χρόνου θα έχουμε το Ευρωπαϊκό Έτος ε, Εθελοντισμού και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν αυτοί οι εθελοντές, υπάρχει η εθελοντική προσφορά και που δημιουργεί μία μη εμπορεύσιμη οικονομία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και αυτές τις οικονομίες που δεν είναι εμπορεύσιμες. Τελευταίο στοιχείο η προσβασιμότητα για όλους. Θέλω να το υπογραμμίσω αυτό. Η κυρία Τρέπελ ε, μίλησε, ε, αναφέρθηκε έτσι τροχάδιν ε, στο θέμα της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία. Ε, τώρα η διαβάθμιση, ναι και αυτό είναι σημαντικό θέμα και το θέμα του κατά πόσο είναι δωρεάν ε, η πρόσβαση και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει οποιοδήποτε σε οποιαδήποτε στιγμή να έχει πρόσβαση στον πολιτισμό. Και τελειώνοντας να πω ότι ο Van Gogh ήταν ένας πολύ απλός αλλά πάρα πολύ μεγάλος καλλιτέχνης ε, και αυτή τη στιγμή στο χρηματιστήριο της τέχνης ε, πουλιούνται τα έργα του σε αστρονομικές τιμές. Όμως στη διάρκεια της ζωής του ο Van δεν μπορούσε να ζήσει από την τέχνη του. Αυτό νομίζω πρέπει να μας απασχολήσει λίγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Περζιά. Να ε, υπογραμμίσω μόνο το εξή. Η αντίληψή για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα. Όχι, όχι, σας λέγω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίθηκε σε αυτό που λέτε εσείς, ότι ο πολιτισμός δεν είναι μόνο εμπόρευμα, είναι και οικονομικό αγαθό όμως. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τη σύμβαση της UNESCO. Δηλαδή ακριβώς αυτό δεν θέλουμε ε, να είναι μόνο αποκλειστικά ε, και μόνο εμπόρευμα ο πολιτισμός. Έχουμε προχωρήσει πιο πέρα από αυτό που ορισμένοι θεωρούν. Και εγώ δεν προέρχομαι από ένα κενό αέρος, γι' αυτό σας τα λέω καμιά φορά έτσι. Ο κύριος Μπόρις, παρακαλώ. E, e, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Τρούιπελ για την έκθεση που μας παρουσίασε και επίσης ε, να αναφερθώ σε ορισμένα στοιχεία της ίδιας εκθέσεως. Πρώτα απ' όλα φαίνεται ότι το Ευρωπαίανα θα πρέπει κατά την άποψή μου να κρατήσει δύο βασικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα να κυδεμονεύσει την, το, το ιδιαίτερα διαφορετικό πολιτιστικό αγαθό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βοηθήσει τις ε, χώρες μέλη που έχουν μείνει λίγο πίσω. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Γαλλίας και θα πρέπει και η Επιτροπή μας εδώ να καλέσει τα κράτη-μέλη να ε, προστατέψουν την ε, πολιτιστική τους κληρονομιά γιατί η φθορά καραδοκεί Επομένως ε, θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή ε, με τοπικούς φορείς, περιφερειακούς φορείς, να σώσουμε έργα τα οποία δημοσιεύτηκαν μετά τον, ε, τον πρώτο ή τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ε, θα ήθελα εγώ να αναφερθώ τώρα και στα θέματα των ταινιών ε, ή των, ε, των ντοκιμοντέρ. Εδώ η ψηφιοποίηση θα πρέπει οπωσδήποτε, η ψηφιοποίηση αυτών των έργων θα πρέπει οπωσδήποτε να μπει στο πρόγραμμα Ευρωπαίανα. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι ε, αποτελούν μέλος, μέρος της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Συνομιλίας και φθύρονται πάρα πολύ εύκολα. Εδώ γίνεται λόγος επίσης για το Google, αλλά έχουμε την Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη από τη μία μεριά, με την εικονογραφία, με τις ε, ταινίες, ε, με τα βιβλία, με εργατέχνης, ε, για τα οποία έχουμε ευθύνη είναι μια πολύ πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια από ότι αυτή του Google. Εγώ πιστεύω ότι για όλα αυτά τα ευρωπαϊκά έργα ε, το Ευρωπαϊκά αποτελεί και μια οικονομική ε, διευθέτηση και να σας εξηγήσω ε, υπάρχουν χώρες ε, πολλές οι οποίες δεν ξέρουν πώς μπορούν να αναμίξουν τον ιδιωτικό τομέα στη διατήρηση της πολιτιστικής ε, κληρονομιάς. Κατά αυτήν την έννοια η Ευρωπαϊκή θα μπορούσε να βοηθήσει πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν δε και να καταγραφούν σε ψηφιακή βάση όλα τα ευρωπαϊκά έργα. Και επομένως θα πρέπει η Ευρωπαϊνα να αποκτήσει και ένα εμπορικό σκέλος, έτσι ώστε όλα τα πνευματικά έργα, μάλλον τα έργα πνευματικής δημιουργίας, να μπορέσουν να ε, ε, μπουν στο, στην Ευρωπαϊκή. Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον θα υπάρξουν συνεταιρισμοί ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Και κατά αυτή την έννοια επίσης λέγω ότι η Ευρωπαϊκή θα πρέπει να ε, λάβει μέτρα έτσι ώστε αυτές οι συμπράξεις να είναι σωστές. Και έτσι βεβαίως όσο γίνεται περισσότερα έργα να μπορέσουν να ψηφιοποιηθούν ε, και να μπουν ε, στην Ευρωπαϊκή. Να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή μπορεί να έχει και εμπορικό χαρακτήρα. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τη συνάδελφο Τρίπελ για την εξαιρετική εργασία που ξεκίνησε. Ζητώ συγγνώμη που ε, άργησα και δεν άκουσα από την αρχή. Ε, έγινε λόγος ε, στον ε, ε, Van Gogh. Ναι, αλλά εδώ θυμόμαστε ότι είχαμε και δολοφονία για, την, για για τα πολιτιστικά θέματα, ας πούμε, Απ' την άλλη πλευρά ε, πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνει όσον αφορά την ε, ε, λογοκρισία. Επίσης, το λογισμικό της Ευρωπαϊνα. Ποιο είναι το λογισμικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και ποια θα είναι η δυνατότητα πρόσβασης. Θα είναι επιγραμμική η πρόσβαση. Με ποιο τρόπο θα, θα γίνεται από άποψη τεχνική. Κυρία Έλγα, mes ce... Έλγα, αγαπητοί συνάδελφοι, λέει η κυρία Μπερνάρ ε, Ατού, ε, του, ευχαριστώ πολύ ε, για την εργασία σου. Θα ήθελα να επισύρω την προσοχή όλων στο θέμα της ψυχής που πρέπει να έχει ο πολιτισμός και δεν θα πρέπει να είμαστε διστακτικοί όσον αφορά τον καθορισμό της ε, ε, περιμέτρου του πολιτισμού. Ε, θα πρέπει να μην ε, ξεχνούμε κανένα έργο ε, και κανένα έργο έστω και αν προέρχεται από πολιτισμούς οι οποίοι θεωρούνται λίγο ε, μακρινότεροι και λίγο δευτερότεροι ενδεχομένως. Δηλαδή θα πρέπει η εργασία των εθνολόγων να ληφθεί υπόψη στην ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής. Ευχαριστώ. Στο Γιάννοφ. Άλλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Τρούπελ. Εγώ θα ήθελα να θίξω μια διαφορετική πτυχή αυτού του θέματος. Εδώ και ένα μήνα ε, ασχολούμαι πολύ εντατικά με την Europeana. Πραγματικά με έχει εκπλήξει το εύρος της και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους Ευρωπαίους. Θα ήθελα να πω λίγα πράγματα σε ό,τι αφορά την οργάνωση αυτού του προγράμματος. η οικονομική, τεχνολογική και ουσιώδης ουσιαστική οργάνωση έχει αποδοθεί στο EDL, μια, ε, ένα ε, Ολλανδικό Ίδρυμα. Μια πρόταση θα ήθελα να κάνω, την οποία βεβαίως θα σας υποβάλω και γραπτός. Σχετίζεται με το γεγονός ότι το Ίδρυμα αυτό έχει πραγματικά κάνει πολύ καλή δουλειά μέχρι τώρα. Βεβαίως πιστεύω ότι είναι επιτέλους ώρα να αναπτύξει και στις 27 χώρες μέλη ε, κλαδιά και διάβλους αυτό το Ίδρυμα. Σημεία επαφής έτσι ώστε να μπορούν όλα αυτά τα σημεία επαφής ενεργά να πιέζουν τις κυβερνήσεις των κρατών μελών ε, για την ε, επιπλέον χρηματοδότηση για τη Ευρωπαϊκή και βεβαίως ε, να πιέζουν και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις των κρατών μελών ώστε να προσελκύσουν και άλλη χρηματοδότηση για το μοναδικό αυτό πρόγραμμα. Επίσης, άλλη μια σημαντική συμβολή θα ήταν η σύμπραξη των εθνικών προσπαθειών έτσι ώστε να υπάρξει μια ενιαία ε, μέθοδος ψηφιοποίησης για να, και να δοθεί και ένα ενιαίο υλικό περιεχόμενο. Εγώ πιστεύω στην περιφερειοποίηση του project αυτού, του προγράμματος αυτού, γιατί θα έφερνε πραγματικά το πρόγραμμα πολύ πιο κοντά στους Ευρωπαίους ε, πολίτες και θα έφερνε αποτελέσματα άμεσα. Κλείνοντας, να πω πως ε, δεν μπορούσα, δεν κατάφερα να βρω στα έγγραφα που έχουμε στα χέρια μας, ίσως να κάνω εγώ βεβαίως λάθος, αλλά δεν κατάφερα να βρω ποιος ελέγχει το Ίδρυμα. Δηλαδή υπάρχει κάποιο σώμα, κάποια αρχή, κάποιο συμβούλιο που εποπτεύει τις δραστηριότητες αυτού του Ιδρύματος. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Νεβεντάλοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα στηρίξω κι εγώ τους ε, υπολείπους. Ε, θα ευχαριστήσω κι εγώ την κυρία Τρούπελ. Είναι εξαιρετική η έκθεσή της. Θα ήθελα να πω κάτι που ήδη υπόθηκε για τους ε, νέους. Εγώ αγοράζω τουλάχιστον 100 βιβλία το χρόνο στην ε, Σλοβακία για να υποστηρίξω τους ε, βιβλιοπόλες στην ε, Σλοβακία. Αλλά δεν έχει ο καθένας αυτή τη δυνατότητα, οπότε αν κάποιος μπει σε μια βιβλιοθήκη στη Σλοβακία μπορεί είτε να πληρώσει μεμονωμένα για ένα βιβλίο είτε να έχει μια συνδρομή ετήσια. Ίσως αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε και για τη Ευρωπαϊκή. Αυτές τις δύο δηλαδή πιθανότητες και αν ας πούμε κάποιος θέλει να, κατεβάσει ε, πορνογραφικό υλικό, ε, αυτό δεν θα πρέπει να το μεταφέρουμε και στην, ε, όταν θέλει κάποιος να κατεβάσει βιβλία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την συνάδελφο Τρούιπελ για την εξαιρετική έκθεσή της. Πρέπει να πω ότι πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο ε, και ιδιαίτερο αλλά και δύσκολο αλλά και δύσκολο ταυτόχρονος. Πρόκειται για μια πρόκληση πάρα πολύ σημαντική. Και παρά τα όσα είπε κάποιος από τους προλαλήσαντες, ε, νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα ε, ε, αποτελεί και έκφραση της εθνικής αλλά και της ευρωπαϊκής ταυτότητας στις οποίες εγώ πιστεύω ακράδαντα. Βεβαίως ε, πρέπει να στηρίξουμε τους δημιουργούς. Βεβαίως ε, θα πρέπει να δούμε αυτό το μεγάλο ζήτημα της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων από τη μία ε, και της οικονομικής διευθέτησης από την άλλη. Ο κύριος Σμιτ μάλιστα ρώτησε προηγουμένως και την κυρία Τρίπελ κάτι που ήθελα να ρωτήσω και εγώ, δηλαδή τι γίνεται σε σχέση με τον προπολογισμό όσον αφορά το πρόγραμμα Ευρωπαϊκά ε, μια και προηγουμένως κάποιος έλεγε ότι θα πρέπει εμείς να διασφαλίσουμε την δωρεάν ε, πρόσβαση. Να πω το εξής, στις ε, πόλεις μας. Ε, όντως ε, έχουμε εμείς κάποιους κανόνες που διευκολύνουν την πρόσβαση και όπως έλεγε και η Στάνης προηγουμένως στις χώρες μας, στις πόλεις μας υπάρχει πάντα η δυνατότητα να πληρώνει κανείς μια εισφορά μηνιαία ή ετήσια και να έχει πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό έργων. Γιατί τι να σας πω τώρα και εντελώς δωρεάν, δηλαδή να έχει κανείς την εντύπωση ότι όλα μπορεί να τα κάνει δωρεάν και όλα θα πρέπει να επιχορηγούνται από το δημόσιο χρήμα, δεν το θεωρώ και απολύτως σωστό. Στις μελέτες όμως που ζητήσαμε ως Επιτροπή υπάρχει μία ε, μελέτη η οποία αφορά ακριβώς ε, την ε, δυνατότητα έβρεσης χρημάτων, πόρων, με κίνων και χορηγών και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί η Ευρωπαϊκή. Δηλαδή θα πρέπει να δημιουργήσουμε την δομή αυτή η οποία οικονομικά θα μπορέσει να στηρίξει το πρόγραμμα το οποίο, ξαναλέω για μία ακόμα φορά, θεωρώ ότι είναι σημαντικό και ουσιώδου σημασίας. Ε, πρέπει να δούμε λοιπόν και τα πρακτικά ζητήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Τούν. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ. Παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή τα όσα είπε η κυρία Τρούπελ. αλλά την έχω ζήσει και σε άλλες επιτροπές ε, με πολύ μεγάλη δέσμευση και στένος υπερασπίζεται αυτό το εγχείρημά της και της εύχομαι κάθε επιτυχία. Υπάρχουν μερικά θέματα τώρα που για μένα ε, εμφανίζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτή η ιστορία με το Google. Εγώ είμαι επιπισμένη ότι όταν κάποιος ε, πιστεύει ε, σε ένα σχέδιο, όταν ε, με σοβαρότητα το προωθεί, μπορεί να έχουμε προώθηση στο διαδίκτυο της λογοτεχνίας με πολιτισμένο τρόπο. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τώρα μονοπόλιο από τις Ηνωμένε Πολιτείες που να περιστέλει τα δικαιώματα των δημιουργών και τα πνευματικά δικαιώματα. Αυτό θα είναι εις βάρος της πολιτιστικής μας και της ιστορικής μας κληρονομιάς και θα αποτελέσει μεγάλο πρόβλημα. Εμείς λοιπόν από την πλευρά μας έχουμε τώρα την ευκαιρία να αντιπαραθέσουμε ε, στην άλλη πλευρά μια διαφορετική αντιμετώπιση και όπως είπε και ο κύριος Σπόρης να προστατεύουμε και τα σύγχρονα έργα Τη σύγχρονη εποχή. Καλή η ψηφιοποίηση, αλλά θα πρέπει να σεβόμαστε τα πνευματικά δικαιώματα σε όλα τα κράτη-μέλη βεβαίω. Αν κατάλαβα καλά, δεν φταίνε οι διαφορές που έχουμε μεταξύ μας για τις καθυστερήσεις και για τις ολιγορίες ε, και τα εμπόδια που γνωρίζει το πρόγραμμα. Ε, μπορεί τα κράτη-μέλη να έχουν διαφορετική νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά δεν είναι πια και τόσο τραγικές ε, οι διαφορές για να μπορούν να καθυστερήσουν, να σταματήσουν ακόμα το εγχείρημα αυτό. Επίσης, ορισμένες χώρες όπως η Γαλλία, για παράδειγμα, έχουν ήδη περάσει στο ψηφιακό σύστημα πολλά έργα, ενώ κάποιες άλλες χώρες πολύ λιγότερα. Θα ήθελα λοιπόν να ενθαρρύνω τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο ενώ νομοθετικό έτσι ώστε να είμαστε εξασφαλισμένοι. Και εμείς και οι δημιουργοί για την προστασία των πνευματικών τους δικαιωμάτων και να μπορέσουμε να στήσουμε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα. Εγώ είμαι από την Κρακοβία. Γνωρίζετε ότι η Κρακοβία είναι η πόλη των ποιητών και πρόσφατα Άκουσα από ποιητές ότι βρίσκουν στο διαδίκτυο ποίηματά τους πολύ κακά μεταφρασμένα. Λοιπόν, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς για την Ευρωπαϊκή να την προετοιμάσουμε και αυτό είναι δουλειά της δικής μας Επιτροπής, να την προωθήσουμε με την αντίστοιχη ενημερωτική εκστρατεία και πληροφόρηση, έτσι ώστε όλα τα κρατη να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια και να προωθήσουν ε, ακόμα περισσότερο την ψηφιοποίηση. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα να πω, κυρία Πρόεδρε, ότι καταλαβαίνω ότι, έχετε, ότι είστε ε, εκπαιδευτικός ε, και φαντάζομαι ότι έχετε μάθει να μιλάτε μπροστά σε τάξη. Πάντως, η παρουσία στην στην ε, Ολομέλεια την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ε, πολύ ικανοποιητική όσο είσαστε και στην ε, Προεδρία. Πάντως πέρα από αυτό, αυτά που είπε η κυρία Τρούπελ ήταν πάρα πολύ σωστά και πολύ σημαντικά ταυτόχρονος και θα αναφερθώ σε ορισμένα. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό, το σημείο κλειδί, είναι το copyright, είναι τα πραγματικά δικαιώματα και η προστασία τους και χαίρομαι πάρα πολύ που ακούστηκε επανειλημμένα ε, το θέμα ε, αυτό. Εμείς έχουμε ε, πριν από 1500 χρόνια στην ιστορία μας μία Μία ιστορία ε, η οποία αφορά ένα πόλεμο που ξεκίνησε ακριβώς ανάμεσα ε, στον ε, Φίνη και στον, σε ένα μοναστήρι, γιατί εκεί είχε ε, γράψει ένα βιβλίο το οποίο το κράτησαν στο μοναστήρι και ο Μεγάλος Βασιλιάς αποφάσισε ότι τελικά θα πρέπει κάθε βιβλίο που θα... του έδωσε δίκιο και είπε ότι κάθε βιβλίο δικό του ε, που θα πουλιέται, τέλος πάντων που θα γράφεται, ε, θα πρέπει να το πληρώνεται και αυτό ονομάστηκε The Battle of the Book, ο, η μάχη του βιβλίου. Ε, και μάλιστα ε, η ιστορία λέει Ε, η ιστορία λέει ότι τότε αποφάσισε να πάει σε πόλεμο και να σκοτώσει όσους ε, και, να ε, εκχριστιανίσει, να προσιλητήσει στον χριστιανισμό όσους είχαν σκοτωθεί στη διάρκεια αυτής της μάχης του βιβλίου. βέβαια η ιστορία δεν μας αναφέρει εάν ε, οποιονδήποτε και στο Independence Party της Ιρλανδίας, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνουμε και από αυτή την ιστορία πόσο παλιά, από πόσο παλιά κρατάει αυτή η μάχη και οποιαδήποτε παραβίαση των πραγματικών δικαιωμάτων στο Google ή οπουδήποτε αλλού είναι ε, κατηγορητέα. Δεύτερον, ε, θα πρέπει να υπάρχει μια, ε, ένας ε, κανόνας κώδικας δεοντολογίας και θα πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το μέλλον μας. Επίσης, η προσβασιμότητα. Ο καθένας από τους πολίτες θα πρέπει να έχει πρόσβαση, αλλά και ο καθένας από τους δημιουργούς θα πρέπει να αμείβεται για την δημιουργία του. Αυτά ήθελα να πω και σε ευχαριστώ κυρία Τρίπελ. Um η κυρία Τρούπελ Τρούπελ έχει ένα πρόβλημα. Πρέπει να φύγει στι 4.30. Έχω τρει ακόμα ομιλητέ. Θα σα παρακαλούσα ένα λεπτό έκαστο και όχι παραπάνω, Αλλιώ δεν θα προλάβει να απαντήσει η κυρία Τρούπε. Ο κύριος Ράτιμο. Ωραία. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο κύριος Βάτιμο, και εγώ βεβαίω θαυμάζω ιδιαίτερα στην εργασία της κυρίας Τρούπελ. Είχα να κάνω δύο-τρεις παρατηρήσεις, ε, οι οποίες ίσως να φανούν και χρήσιμες. Πρώτη παρατήρηση. Προτείνεται, προβλέπεται κάποια χρονική διαβάθμιση στην ε, πραγματοποίηση του προγράμματος, γιατί φοβούμε το εξής η ιδέα της ψηφιοποίησης των πάντων φοβούμε ότι τελικά θα επιβραδύνει ιδιαίτερο στην εργασία μας. Ας πούμε μόνο στην κινηματογραφία ή στη μουσική γιατί το θέμα του downloading της ε, μουσικής είναι το πιο σημαντικό και εκεί βασίζονται και αυτοί οι Σουηδοί πειρατές. Γιατί δεν διάβασα τίποτα για βιβλία, φαίνεται ότι δεν τους ενδιαφέρουν τα βιβλία, κανείς δεν ενδιαφέρεται για τα βιβλία. Όλα τα παιδιά κάνουν, ε, κατεβάζουν ε, μουσική. Θα μπορούσαμε λοιπόν να προτείνουμε ένα τρόπο χρονικής διαβάθμισης. Ας πούμε, αν ξεκινούσαμε από τα βιβλία. Πολλά από τα προβλήματα δεν θα παρουσιάζονται για τα βιβλία. Γιατί σε, όλες ε, τις, ε, σε όλους τους εκδοτικούς οίκους κάποια στιγμή εκπίπτει ο χρόνος ε, των πνευματικών δικαιωμάτων και επομένως ίσως θα ήταν πιο εύκολο να ξεκινήσουμε από εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχηθώ και εγώ συγχαρητήρια στην κυρία Τρούπελ για την έκθεσή της. Και για να εξοικονομήσουμε χρόνο, δεν θέλω να επαναλάβω όσα είπαν οι προλαλήσαντες, μόνο το εξής. η Ευρωπαϊκή είναι άμεσος ανταγωνισμός για την Google. Γιατί αν συμβαίνει αυτό, τότε ε, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα για μας. Την Ευρωπαϊκή θα έπρεπε να τη δημιουργήσουμε ακόμα και αν δεν υπήρχε το Google. Το, η πολιτιστική κληρονομία στην Ευρώπη είναι δημόσιο αγαθό. Όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτήν. Αν όμως το εγχείρημα αυτό βασιστεί σε ιδιώτη, φοβάμαι ότι θα έχει βραχή βίο. Οι πηγές χρηματοδότησης είναι πολύ σημαντικές και ο ιδιώτης να είναι ένα μόνο τμήμα. Ε, η κυρία Κάμερα, πάρα πολύ σύντομα και να τελειώσουμε. Συγγνώμη, κάτι τέλειωσα προηγουμένως για το δωρεάν, δεν θα ξαναπώ τίποτα, λέει η κυρία Κάμερβερτ. Η κυρία Τρούπελ στην έκθεσή της μίλησε για εταιρείες συλλογική εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων πνευματικής ε, ιδιοκτησίας και είναι και θέματα σημαντικά αυτά για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Από άλλε συζητήσει όμω γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το καιρό δυσκολεύει πάρα πολύ ε, τη ζωή των εταιριών που ήδη υπάρχουν γιατί του κατατάσσει στον κλάδο του ανταγωνισμού και τους υποπτεύεται τους άνθρωπους αυτούς για στρέβλωση, λέει, του ανταγωνισμού. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να μας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό, πώς μπορεί να λυθεί και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή. Okay. Äh, Ωραία. Οπότε να δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν, αν μπορείτε να είστε και σύντομος, γιατί η κυρία Τρόπελ μετά θέλει να πάρει το λόγο, να απαντήσει και πρέπει και να φύγει. Καταρχάς θα ήθελα συγχαρώ την κυρία Τρούπελ και συγχαρητήρια κυρία Πρόεδρε και ε, κύριοι βουλευτές για τον ενθουσιασμό που επιδεικνύεται για την Ευρωπαϊκή. Η έκθεση κυρία Στρούπελ είναι πραγματικά καταπληκτική. Ε, έχει εγγίξει ε, όλα τα θέματα και τα σημαντικότερα βέβαια πάντα. Από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούμε ότι είναι πολύ φιλόδοξο αυτό το πρόγραμμα και η θύρα ο ιστότοπος είναι πολύ σημαντικός ε, και βιτρίνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι μόνο η κορφή του παγόβουνου. Δείχνει τις προσπάθειες που έχουν κάνει τα κράτη-μέλη και οι πολιτιστικοί φορείς για την ψηφιοποίηση. Θα πρέπει λοιπόν επίλημα αυτή η δικτυακή να ενισχυθεί από πολλούς φορείς. Υπάρχουν μερικά σημεία τα οποία δεν ακούστηκαν και θα ήθελα να τονίσω, αν μου επιτρέπετε. Πρώτον, τα λεγόμενα ορφανά έργα και ο κατεπήγων για τη λύση τους, ειδικά όταν μιλάμε για οπτικοακουστικά ντοκιμαντέρ είναι τεράστιος ο όγκος. Οι ταινιοθήκες στην Ευρώπη μας είπαν ότι έχουν 50.000 ταινίες που μπορούν να ταξινομηθούν ως ε, ορφανά έργα. Είναι τεράστιος όγκος, 50.000. Το δεύτερο θέμα είναι τα λεγόμενα έργα που προστατεύονται από πνευματική ιδιοκτησία. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή και στα μεγάλα πολιτιστικά σχέδια εθνικών βιβλιοθηκών βλέπουμε πολλά έργα που είναι ε, δημοσίες ε, χρήσεως και πολύ λίγα που προστατεύονται από ε, πνευματικά δικαιώματα. Και πώς θα λυθεί αυτό για να μην έχουμε μαύρη τρύπα, όπως είπατε, για τον 20ο-21ο αιώνα, θα πρέπει να συνεννοηθούμε με τους συντάκτες, με τους εκδότες, ε, για να συνεργαστούμε, να περάσουν όλα αυτά σε ψηφιακό περιβάλλον. Τι χρειάζεται εδώ πέρα. Εδώ χρειάζεται ε, οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων να έρθουν σε συμφωνία μαζί μας και με έναν τρόπο εύκολο να διαπραγματευτούμε, να ξέρουμε ποιοι είναι οι δημιουργοί, με απλό τρόπο για να προχωρήσουμε. Ένα δεύτερο θέμα που μας ανησυχεί και δεν έφυγε εδώ είναι ότι υπάρχουν μερικές συμφωνίες σε εθνικό επίπεδο μεταξύ πολιτιστικών φορέων, ε, εκδοτών και δημιουργών, συγγραφέων που μπορούν να μπουν μεν τα έγγραφα του στο ίντερνετ, αλλά περιορίζεται η πρόσβαση μόνο για την εθνική επικράτεια. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό θα ήταν ολέθριο. Εάν όλες αυτές οι προσπάθειες ψηφιοποίησης καταλήξουν σε σιλό ε, κατακαιρματισμένα και ε, κλειστά ε, σε κάθε χώρα. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις ένα πάροχο στην Ολλανδία για να μπει στο site της Ολλανδίας και μετά στη Γερμανία το ίδιο κτλ. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθούν. Την Παρασκευή συνεδρίασαν οι Υπουργοί Πολιτισμού και ήταν πολύ ενθουσιώδη τα κράτη-μέλη και αυτό με φέρνει στο μέλλον, είναι νέα πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την Παρασκευή έχουμε νέα επίτροπο για την ψηφιακή ατζέντα και έρχεται σε πολύ κατάλληλη χρονική στιγμή θαυμάσει η έκθεσή σας για να ε, συνεργαστούμε την κυρία Κρούς και την ψηφιακή ατζέντα. Όλοι λοιπόν οι φορείς, ε, οι φορείς του διαδικτύου, οι εκδότες, οι συγγραφείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να πετύχουμε το μεγάλο μας στόχο που δεν είναι άλλος παρά η ευρωπαϊκή μας πολιτιστική κληρονομιά να είναι προσβάσιμη σε όλους μέσω του διαδικτύου με τρόπο εύκολο και πλήρη. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρο. ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέλφους για τα σχόλιά τους, για την κριτική τους, ε, για ε, όλα τα έγγραφα που μου έδωσαν για, την προετοιμασία της έκθεσης. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Καταρχήν, η Europeana θέλω να είναι ένα project το οποίο θα αφορά την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Και αυτό θα το κάναμε ούτως ή άλλως, ανεξαρτήτως αν υπήρχε δηλαδή το Google ή όχι. Το Google τώρα υπάρχει, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς κινούμαστε στον πραγματικό κόσμο μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Φυσικά η Ευρωπαϊκή είναι ένα θέμα, το οποίο, ένα project το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και τα επιχειρήματα προς αυτό ακούστηκαν εδώ. Γιατί δηλαδή είναι σημαντικό και κεντρικό σημείο, κεντρικό πρόγραμμα για την Ευρώπη. Δεύτερη παρατήρηση, όταν μιλούμε για όλη αυτή την ε, ε, το θέμα των, ε, της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, θέλω να βρούμε συμβιβασμούς με, με τους οίκους, με τους κατόχους των δικαιωμάτων, με τους συγγραφείς, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο το περιεχόμενο αυτό, γιατί αυτό σε κάθε περίπτωση ε, είναι σημαντικό. Ε, δεν, όταν δεν μιλούμε για, την, ε, για, το, για, το, για θέματα copyright, αυτό δεν σημαίνει ότι τα πάντα θα είναι δωρεάν. Πρέπει λοιπόν να ε, προσπαθήσουμε. παρόλα όλα αυτά, συμφωνώ ότι πρέπει να είναι ένα ελεύθερο project το οποίο να χρηματοδοτείται και να είναι προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες, ακόμη και σε άτομα με αναπηρία και εκεί θα πρέπει να υπάρξουν ε, κάποιες διασαφηνήσεις και ως προς το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων. Είναι πολιτικό πρόγραμμα, αλλά δεν ε, σημαίνει ότι όλα θα είναι δωρεάν, γιατί όντως και οι συγγραφείς ε, και οι δημιουργοί θα πρέπει να λαμβάνουν κάτι ως αντιστάθμισμα για τα έργα τους τα οποία προστατεύονται. Δεν είναι δηλαδή απλώς ένα μοντέλο που λειτουργεί χωρίς καμία πληρωμή ως προς το περιεχόμενο που, που διαθέτει. Τώρα για το θέμα της εκστρατεία, της χρηματοδότησης ε, του προγράμματος αυτού καθ' αυτού. Ε, θα το ήθελα και θα προσπαθήσω, το έκανα και την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο όταν, την, όταν είχαμε την προφορική ερώτηση για το Google, ε, θα ήθελα όπως είπα το κονδύλι να βγει από το πρόγραμμα της Λισαβόνας για την Ευρωπαϊκή, γιατί αυτό είναι πραγματικά αποφασιστική σημασία ε, θέμα για, την, ε, για τον εξυγχρονισμό και του πολιτισμού και της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό, κύριε Μάρτιν, δεν θεωρώ όπως και εσείς, ότι δεν είναι, ότι είναι καλό ε, έτσι, να μπαζεύουμε από εδώ και από εκεί και να βάζουμε, τα βάζουμε στη Ευρωπαϊκή Πρέπει να υπάρξει μια αναβαρχίδα που να προκύπτει από την ε, Λισαβόνα. Και αυτό θα προσπαθήσω να το προωθήσω. Πρέπει να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο και ο δικός μου πολιτικός στόχος είναι να, γίνει, να είναι σαφώς, να είναι ορατό αυτό και σαφές. Ε, για το e-content plus Έχουμε ένα χρονικό ορίζοντα 2009-2011, ε, συγγνώμη, ένα κονδύλι 2,6 εκατομμύρια ευρώ. τα κράτη-μέλη και, διάφορα, και τα διάφορα ιδρύματα τα πολιτιστικά θα πρέπει να εμπλακούν ακόμη και αν δεν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε πολιτικό επίπεδο γι' αυτό. Τώρα, για την ιδιωτική χρηματοδότηση θα μπορούσαμε να την, θα μπορούσαμε να την δεχτούμε. Θα ήταν σημαντικό όμως το μεγάλο κονδύλι να προέρχεται από, την, από το δημόσιο τομέα. Αλλά επίσης σωστό θεωρώ είναι ότι θα πρέπει να πληρώνονται και οι πνευματικές προσφορές, η δημιουργία ο πολιτισμός και το, και το υλικό έχει, και το πνευματικό υλικό, το δημιουργικό υλικό είναι όντως εμπόρευμα το οποίο πρέπει να φανεί γιατί πρέπει να φανεί τι, τι παράγουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πρέπει να ζήσουν από αυτό. Πρέπει να μπορούν και οι κινηματογραφιστές και οι συγγραφείς να ζουν από τα έργα τους. Δεν προσπαθούμε να τους καταστρέψουμε στον ψηφιακό κόσμο. Ταυτόχρονα όμως ο πολιτισμός είναι και κάτι παραπάνω από εμπόρευμα. Είναι ένας φορέας α, σημασίας λόγου. Αυτό το έχουμε πετύχει και εμείς όταν είχαμε τη σύμβαση της, της UNESCO επιμείναμε στο να και αντιταχθήκαμε στην, στην UNESCO. Αυτή η εξαρτία τώρα που σας ανέφερα για, την, για το Joint Europeana. Ε, δημόσια χρηματοδότηση. Αλλά θα πρέπει να δεχτούμε και την ε, χρηματοδότηση από ιδιωτικούς φορείς Αν μπορέσουμε να τα καταφέρουμε δηλαδή ε, χρηματοδότηση από τέτοια ιδρύματα, φυσικά θα ήταν ε, καλό. Και αν σκεφτούμε και τους νέους και πως μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά τους με άλλα είδη διαφήμιση, εγώ θα ήμουν η τελευταία που θα λέγει όχι. Αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που είπε η κυρία Κάμερ Εύερτ. Όντω η διαφήμιση δεν θα πρέπει να γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται για τον Google και στην Europeana. Τώρα, για το περιεχόμενο, το, είπε, το ρώτησαν αρκετοί συνάδελφοι για τι βιβλιοθήκε που θα ψηφιοποιηθούν και θα, και θα διαβιβαστούν τα περιεχόμενά τους και τι περιεχόμενο θα υπάρχει εκεί. Και φυσικά θα πρέπει αυτό το περιεχόμενο να, έχει υψηλή, να είναι υψηλή ποιότητα. Επίση το open software, αν αυτό θα λειτουργήσει για την Europeana. Εγώ, από όσο ξέρω, θα έχουν δική τους πλατφόρμα, θα έχει δική τους πλατφόρμα η Europeana για το λογισμικό. Δεν θα είναι με open software. Θα έχει δικό τους μοντέλο. Αλλά εντάξει, αυτό μπορούν να μας το λύσουν και οι εμπειρογνώμονες και αυτοί που θα είναι υπεύθυνοι, οι διευθυντές δηλαδή, με τους συνεργάτες τους που θα είναι υπεύθυνοι για την, ε, για την θα μας βοηθήσουν περαιτέρω επ' αυτού. Τελευταία παρατήρηση. Κατέστη σαφές, ε, παρόλο που έχουμε, θα δούμε και τις ε, τροπολογίες που υπάρχουν, έχω την εντύπωση ότι σε όλη την ομάδα υπάρχει μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον για, το, για να προωθηθεί η Ευρωπαϊκή να εξελιχθεί και γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Χέλγα. Όντω, έχουμε την εντύπωση ότι πραγματικά εργαζόμαστε από κοινού για ένα κοινό πρόγραμμα. Ο κύριο Καβαντά πραγματικά με εντυπωσίασε με αυτό που είπε. Όλα όσα συλλέγουμε εδώ παράγονται με τελείως διαφορετικό τρόπο και θα παράγονται με τελείως διαφορετικό τρόπο όταν, ε, δεν θα, όταν θα αλλάξουν τελείως τα πράγματα στο ψηφιακό περιβάλλον. Κάποτε είχαμε και εμείς στον καιρό μου ένα βίντεο, μετά έγινε DVD. Ε, οι, οι δυνατότητες που έχουμε τώρα είναι τεράστιες και ούτε καν α, τις ξέραμε όταν ήταν ε, ο καιρός του βίντεο κάποτε. Οπότε ε, ακόμα όσο θα εξελίσσονται οι ε, τεχνολογίες τα πράγματα θα είναι, θα είναι πολύ διαφορετικά. Αλλά ακόμη και τότε αυτά τα σημερινά που είναι υψηλής τεχνολογίας μέσα θα είναι παλαιωμένα. Πραγματικά λοιπόν πρέπει να καταλήξουμε σε ένα καλό ποιοτικό αποτέλεσμα και γι' αυτό χρειαζόμαστε και την συνεργασία των κρατών μελών. Εγώ είμαι σίγουρη ότι ακριβώς αυτή η συζήτηση για το Google γίνεται και σε πολλά κράτη-μέλη, από τους εθνικούς βουλευτές, συζητιέται το θέμα αυτό, για να μπορέσουμε να, να, να διασφαλίσουμε την ευρωπαϊκή διαφορετικότητα. Λοιπόν, ε, τροπολογίες, προθεσμία για τροπολογίες. Πότε είναι? Στις 12. Στις 8. Την επόμενη εβδομάδα, 8 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι. 8 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Και στις 26 θα την κάνουμε τη συνεδρίαση ή όχι, 26 Ιανουαρίου. Θα πρέπει να ψηφίσουμε για την Ευρωπαϊκή. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με την Ολομέλεια, τη μήνυ Ολομέλεια για τους επιτρόπους και τις ε, ακροάσεις. Θα το δούμε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 8 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι, ε, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Πάμε στο σημείο 5. Ε, διάλογος πανεπιστημίων επιχειρήσεων, μια νέα εταιρική σχέση για τον εξυγχρονισμό των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Στις 2 Σεπτεμβρίου ο συνάδελφος Σμιτ ήταν ε, ορίστηκε εισηγητής για το θέμα αυτό. 13 Οκτωβρίου η Επιτροπή Ήτρε ζήτησε να ε, συμμετάσχει στο με το δυνάμει του σημείου 50 του ιστορικού κανονισμού. Ε, έχουμε λοιπόν ένα κοινό χρονοδιάγραμμα. Ο κύριο Σμιτ νομίζω το έχει κάνει όμως όλα αυτά. Θα δώσω κατευθείαν το λόγο στον κύριο Σμιτ ε, για να μας πει τι έχει γίνει μέχρι στιγμή και τι γίνεται και με την συνεργασία με την Επιτροπή Ήτρε. Παρακαλώ Παλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την έκθεση αυτή με τον κύριο Σκούρια. Όσο προετοιμάζομαι και διαβάζω και ενημερώνομαι, βλέπω πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Ρίτα Σουάρες για τη βοήθειά της, που πραγματικά ήταν πολύτιμη στην υποστήριξη της. Έχουμε τις διάφορες ανακοινώσεις τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις μελετήσαμε και ε, επίση μελετήσαμε και το υπόλοιπο υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας. Στενότερη συνεργασία επιχειρήσεων και πανεπιστημίων είναι από τα βασικότερα στοιχεία και τα σημαντικότερα της στρατηγικής της Λισαβόνας. Και αυτό εξυπηρετεί δύο στόχους. Ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης αφενός και αφετέρου εξυγχρονισμό των πανεπιστημίων. Για τους νέους θα πρέπει να είναι ο στόχος ως εξής όλοι οι φοιτητέ και όλοι οι σπουδαστέ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι και με πρακτική εμπειρία και με πρακτική γνώση, γνώση ε, όταν παίρνουν το δίπλωμά τους, να έχουν και επαφή με τις επιχειρήσεις για να μπορούν να βρουν καλύτερα δουλειά στη συνέχεια. Και για τους διδάσκοντες είναι πολύ σημαντικό αυτό για να ξέρουν ποιες είναι οι ανάγκες ε, της αγοράς εργασίας, να τις σταθμίζουν και να εκπαιδεύουν ανάλογα και τους φοιτητές τους. Να είναι ανοιχτά λοιπόν τα πανεπιστήμια ε, στις επιχειρήσεις, ε, στον οικονομικό κόσμο, αλλιώς Ε, ε, θα υπάρχουν ε, προβλήματα. Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις χρειάζονται και τους ακαδημαϊκούς εμπειρογνώμονες. Τα αποτελέσματα βεβαίως δεν είναι πρόθεσμα αλλά εδώ θα πρέπει να υποστηρίξουμε κάθε προσπάθεια που θα βγάλει την Ευρώπη από την κρίση και θα μειώσει την ανεργία. Το έγγραφο που έχουμε εδώ είναι μόνο έγγραφο εργασίας, έτσι, και ομιλεί για τις προτεραιότητες που θεωρώ εγώ σημαντικότερες. Μεταξύ των προτεραιοτήτων αυτών θα ήθελα να σας αναφέρω τα εξής. Το πλαίσιο του διαλόγου θα πρέπει να είναι σαφές και τα θέματα του διαλόγου, αλλά επίσης και οι συμμετέχοντες στο διάλογο αυτό. Το θέμα είναι τώρα τι διάλογος θα είναι, θα είναι διμερής, μήπως να καλέσουμε και τις κυβερνήσεις. να μην είναι μόνο διμερείς δηλαδή επιχειρήσεις και πανεπιστήμια, αλλά να διευκολύνεται το όλο εγχείρημα από τις κυβερνήσεις. Και ποιος να είναι ο στόχος. Έχουν γίνει πολλές διασκέψεις, συζητήσεις, ανταλλαγές απόψεων. Ε, κάποια στιγμή φτάνει η ώρα των αποτελεσμάτων, των απλών, απτών και χειροπιαστών. Και γι' αυτό θα ήθελα να μου δώσετε και συμβουλές και να μου κάνετε και παρατηρήσεις. Άλλο θέμα, πώς συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. που δεν έχουν για πολλούς οικονομικούς πόρους και δεν έχουν και μεγάλο μερίδιο από την πίτα. Λοιπόν, ε, θα πρέπει επίσης να κοιτάξουμε τι γίνεται με τα μέλη της Euronest ε, της, ε, ή της Ένωσης ε, της Μεσογείου ή υποψήφιες χώρες, πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τις γειτονικές μας χώρες με άλλα λόγια. Εγώ είχα ένα διάλογο με την επικεφαλή στη Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Κατάρτισης και δηλώνει πρόθυμη να συνεργαστεί μαζί μας. Άλλη πτυχή είναι επαγγελματική κατάρτιση και τα ΤΕΙ, ε, ας πούμε, οι σχολές, τεχνικές σχολές μέσης εκπαιδεύσεως για να μπορούν να συνεχίσουν τις τεχνικές σπουδές τους και τις επαγγελματικές τους. Δεν θα πρέπει εδώ να δημιουργούνται τεχνητά εμπόδια για τους σπουδαστές επειδή έχουν τελειώσει λάθος σχολείο, για παράδειγμα, τεχνική σχολή. Ε, άλλο θέμα παρακολούθηση και συνέχεια να δίνεται από τα πανεπιστήμια για να κοιτούν τα πανεπιστήμια και να γνωρίζουν ποια είναι η σταδιοδρομία που ακολουθούν οι φοιτητέ τους και να τα καταγράφουν και να, παρακολουθούν, να ξέρουν τα πανεπιστήμια τι πτυχίου βγάζουν και τι απασχόληση έχουν αυτή στη συνέχεια στη ζωή τους. Γιατί ε, από μια πρώτη γεύση που πήρα δεν έχουν ιδέα τα πανεπιστήμια που καταλήγουν οι πτυχιούχοι τους και τελικά που εργάζονται. Θα ήθελα επίσης να σας επιστήσω την προσοχή ε, στο εξή γεγονό. Εμείς έχουμε ξεκινήσει ακρόαση με τίτλο «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια Προκλήσεις και Απαντήσεις» και απαιτήσει. στι 26 Ιανουαρίου θα γίνει ευθεκρόση και μπορείτε να κάνετε προτάσει στη γραμματεία για ποιου εμπειρογνωμόνε θέλετε να καλέσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί πρόεδρε, περιμένω να ακούσω τι ιδέε σα τα σχόλιά σα για να εμπλουτίσουμε από κοινού την έκθεση αυτή και τη συνεργασία. Και είμαι πεπισμένο ότι, ελπίζω μη τι άλλο, η έκθεση αυτή θα βοηθήσει και να πετύχουμε του βασικού μα στόχου. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάλι. Ο κύριος Λόραγκαρτ. Er Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, γιατί είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι το συζητούμε εδώ και λίγο χρόνο. Δεν είναι εντελώς καινούριο θέμα. Και η άποψή μου είναι ότι πολλά λόγια, αλλά λίγα εξειδικευμένα λόγια και επομένως νομίζω ότι πρέπει λίγο να κινηθούμε τώρα και συμφωνούμε με τον κύριο Σμιτ ότι θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητες στο ζήτημα για να ξεφύγουμε και από την κρίση. Το ζήτημα είναι με ποιο τρόπο. Θα ήθελα λοιπόν να δείξω κάποια συγκεκριμένα θέματα, έτσι σαν τροφή προς σκέψη για τον κύριο Σμιτ. Συμφωνώ με αυτά που αναφέρει στο ανακοινωθέν ε, η Επιτροπή. Αναφέρεται σε έξι θέματα, εγώ θα μιλήσω για δύο από αυτά. Το πρώτο, επί του οποίου πρέπει να επικεντρωθούμε, έχει να κάνει με τα προγράμματα και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να έχουμε διατομιακή προσέγγιση έτσι ώστε όσοι βγαίνουν από τα πανεπιστήμια να ξέρουν, να έχουν ήδη σχέση με την αγορά ε, εργασίας, την καινοτομία και την έρευνα. Det giver sig selv, øh, skulle man synes, det er faktisk ikke tilfældet i dag. Όσον αφορά τώρα τα πανεπιστήμια, εγώ το είδα και από μόνος μου, από τη δικιά μου εμπειρία. Ξέρετε, είναι δύσκολη η επαφή ανάμεσα στο πανεπιστήμιο και την αγορά εργασίας, γιατί ε, οι δύο πλευρές μιλούν διαφορετική γλώσσα, έχουν διαφορετική κουλτούρα και επομένως ε, το διακύβευμα, η πρόκληση αν θέλετε, είναι αυτή ακριβώς, το να βρούμε μια κοινή γλώσσα ανάμεσα στον κόσμο του Πανεπιστημίου και τον κόσμο της αγοράς και αυτό δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Συμφωνώ με τον κύριο Σμιτ ότι η κατάρτιση, η διαβίου κατάρτιση, ε, η συνεχής μαθητεία οπωσδήποτε θα πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών των πανεπιστημίων έτσι ώστε να έχουμε μια πραγματικά ε, διαρκή κατάρτιση στα πανεπιστήμια. Τρίτον, έλλειψη μηχανικών, έλλειψη ενδιαφερομένων για τις φυσικές σπουδές ε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα στη Δανία. Εδώ και τρία-τέσσερα χρόνια προσπαθούμε να βρούμε μια λύση στο πρόβλημα αυτό, αλλά παρά τι ε, πρωτοβουλίε, ε, παρά τι υποσχέσει και τα μεγάλα λόγια δεν έχουμε βρει ακόμα λύση. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ενδιαφέρον για τις ε, φυσικές επιστήμες και ε, βεβαίως όταν φτάσει κανείς στο πανεπιστήμιο είναι ήδη αργά να του πεις τώρα γίνε, επίλεξε αυτή την κατεύθυνση και γίνε μηχανικός. Ας πούμε. Πρέπει η δουλειά να γίνει πιο πριν. Επίσης, ε, θα έλεγα προηγουμένως ότι πρέπει να δημιουργήσουμε, ε, να βρούμε μια κοινή γλώσσα. Λέω τώρα ότι πρέπει να δημιουργήσουμε διάβλους επικοινωνίας. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και έπειτα η έρευνα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και η έρευνα θα πρέπει να δημιουργήσει περάσματα και γέφυρες. όταν είμαστε σε μία επιχείρηση θα πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθούμε και σπουδές ε, στο πανεπιστήμιο και αυτό θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από τα πανεπιστήμια, από τους αρμόδιους ε, υπουργούς ε, υγείας έτσι ώστε να δημιουργήσουμε κοινέ πραγματικά προσπάθειες και έτσι ώστε άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν να μπορούν να σπουδάζουν ταυτόχρονα και μάλιστα να μπορούν να σπουδάζουν και στο εξωτερικό. Ε, πρέπει να σας πω ότι στην Δανία δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα όπου το κράτος έδινε 60.000 ευρώ επιδότηση σε κάποιες επιχειρήσεις έτσι ώστε να δώσουν τη δυνατότητα τρίχρονης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ε, ε, στους υπαλλήλους τους, στους εργαζομένους τους και αυτό είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να μάθουμε και από το παρελθόν. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να έχουμε τρομερές νέες ιδέες. Υπάρχουν οι ιδέες, απλώς πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε. Ε, πρέπει να βρούμε και χρήματα βεβαίως, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν τα χρήματα στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Επομένως, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο με αυτό που σας ανέφερα στη Δανία. Ευχαριστώ, η κυρία ε, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Σμιτ. Έχετε κάνει καμία έρευνα στα πανεπιστήμια που έχουν θεωρητικές σπουδές υπάρχει συνεργασία με τις επιχειρήσεις και πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ας πούμε όταν κάποιος σπουδάζει φιλολογία, μια ξένη γλώσσα, ποιες είναι οι επιχειρήσεις, ποια είναι η αγορά εργασίας, οι εταιρείε μεταφραστών, εντάξει. Από εκεί και πέρα ποιος άλλος μπορεί να ενδιαφέρεται. Γιατί στη δική μου χώρα είναι υποχρεωτική άσκηση ε, το πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια της φίτησης ο καθένας στον τομέα του. Ε, και υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός εβδομάδων για πρακτική άσκηση που είναι υποχρεωτική για να μπορεί κανείς να πάρει πτυχίο και να του δώσουν και ένα πιστοποιητικό ότι έχει εμπειρία πρακτική. Θα μπορούσε ίσως και αυτό να είναι μια πρόταση, μια ιδέα, δεν ξέρω αν το σκεφτούμε, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων. Ας πούμε, στη χώρα μου όλοι θέλουν να σπουδάσουν νομικά. Πολυτεχνείο κανείς. Ε, αυτό είναι ένα πρόβλημα σε όλη την Ένωση νομίζω. Υπάρχουν κάποιες σχολές που δεν εμφανίζουν ενδιαφέρον φοιτητές. Θα μπορούσαμε λοιπόν να υποστηρίξουμε αυτή την πρόταση και να το κοιτάξουμε και αυτό Ευχαριστώ. Κύριος Ρέπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξαιρετική ήταν σήμερα η ημέρα μας. Η Ευρωπαϊκή πραγματικά είναι το απάβγασμα του ήθους της Ευρώπης. Έχουν γίνει πάρα πολλά, αλλά το σημαντικό είναι πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά που έχουν, ε, που έχουν γίνει και σε ό,τι αφορά τον ακαδημαϊκό κόσμο και σε ό,τι αφορά τον επιχειρηματικό κόσμο. Χρειαζόμαστε τον πολιτισμό. Και φυσικά πρέπει και ο οικονομικός τομέας να έχει μέλλον. Εγώ είμαι ο σκιώδης εισηγητής ε, για το θέμα αυτό πρώτη φορά και συμφωνώ ε, με αυτά που αναφέρει η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της. Ο κύριος Σμιτ επίσης ανέφερε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και ως Φιλανδός, από την αρχή του επόμενου ε, ε, έτους πρέπει να σας πω ότι εμείς θα έχουμε ένα νέο πανεπιστήμιο ε, με, που θα γίνει μια σύμπραξη των οικονομικών σχολών και των τεχνικών σχολών, καθώς επίσης και, του, ε, ε, και της σχολής καλών τεχνών και βιομηχανικού σχεδιασμού. Οπότε κάνουμε ό,τι μπορούμε, βλέπετε, για τον διάλογο μεταξύ του επιχειρηματικού και του ακαδημαϊκού κόσμου αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει βεβαίω να επεκταθεί και περισσότερο σε άλλου τομεί της κοινωνία για να μπορέσει να εφαρμοστεί και να αφορά όλους τους εμπλεκόμενου φορείς ε, και τις ε, ε, ενώσει της αγορά εργασία, άλλου φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, δημόσιου φορείς. Κατά αυτόν τον τρόπο, πιστεύω ότι η διεύρυνση του διαλόγου είναι πολύ σημαντική Ε, πρόσφατα έγινε μια, ε, μια παρουσίαση για την επιχειρηματικότητα ε, στην Κομισιόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ακούστηκαν απόψεις που αφορούν την Κίνα στην Ουψάλα. Όταν ρωτήσει κανείς τους ε, ε, φοιτητές, τους Κινέζους φοιτητές ε, πόσοι που σπουδάζουν διοίκηση επιχειρήσεων, πόσοι θέλετε να γίνετε επιχειρηματίες, όλοι σήκωσαν το χέρι τους. Στη Σουηδία και στη Φιλανδία 5% σήκωνε το χέρι του από τους φοιτητές που θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες. Οπότε αυτό μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει σύγκληση μεταξύ ακαδημαϊκού κόσμου και επιχειρηματικού πνεύματος. Αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουμε σοβαρά υπόψη μας. Ευχαριστώ. Κύριε Κέλλη. Thank you very much. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι πολύ με ευχαρίστησαν ε, όλα αυτά τα οποία σαφώς ανέφερε ο κύριος Σμιτ. Νομίζω ότι μπορώ να συμφωνήσω απολύτως με όλα αυτά που είπε ε, και σε σχέση με το, αυτό που ανέφερε ότι θα πρέπει οι επιχειρηματίες και τα πανεπιστήμια να συνδεθούν μέχρι τώρα. Για πολλά χρόνια τα πανεπιστήμια έζησαν μέσα σε αλαβάστρινους ε, πύργους ε, και έβγαιναν τα παιδιά από το πανεπιστήμιο με κάποιες γνώσεις αλλά χωρίς καμία εμπειρία, χωρίς ε, τίποτα απτό. Βέβαια τα πράγματα άλλαξαν ε, ε, ε, φέτος, συγγνώμη, τον τελευταίο καιρό. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αφενός να είναι συνδεδεμένοι όταν σπουδάζουν με την αγορά εργασίας για να ξέρουν τι θα κάνουν και μετά και αφετέρου επιχειρηματίες οι οποίοι να είναι μορφωμένοι και να μπορούν να προχωρήσουν σωστά. Αυτό που μας ενδιαφέρει βεβαίως είναι να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και να διερευνήσουμε τον τομέα της ανάπτυξης και της ε, έρευνας και μία μελέτη η οποία έγινε πρόσφατα σε μεγάλο πανεπιστήμιο έδειξε ακριβώς ότι η ακολουθητέα οδός είναι αυτή που καταδεικνύει και ο κύριος ε, Σμιτ. Ε, είναι πάρα πολλά τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να απασχολήσουν πλέον και τα πανεπιστήμια, η τεχνογνωσία, η πραγματογνωμοσύνη όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές, όσον αφορά τις νέες συνθήκες διαβίωσης. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι, είτε είναι στα πανεπιστήμια, είτε είναι στην πραγματική ζωή. Ε, και κύριε Σμιτ, πολύ καλή δουλειά να ε, συνεχίσετε. Ο κύριος Κουρία. μια και ο κύριος Σμίτε μας ζήτησε και πρακτικές συμβουλές και βεβαίως εδώ να τον ευχαριστήσω πρώτα για την εργασία που έκανε η οποία έδειξε ήταν άξιος της εμπιστοσύνης που του δείξαμε. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε κάποιες εμπειρίες τις οποίες υλοποίησε ε, το Υπουργείο Νεότητας της Ιταλίας. Πρώτον, δημιούργησε ένα είδος μηνιαίου κάμπους ε, όπου 100 φοιτητές οι οποίοι αξιοκρατικά έχουν επιλεγεί από τα Πανεπιστήμια της Ρώμης για μία ή μία μισή εβδομάδα έρχονται να συναντήσουν ε, μεγάλες ευρωπαϊκές ή πολυεθνικές εταιρείες, Fiat, Microsoft κλπ έτσι ώστε να τους ε, υποβάλουν ε, τα βιογραφικά τους, να συζητήσουν τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων και όλα αυτά υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου έτσι ώστε να μην αφήσουμε τους νέους μόνους τους ε, στην αγορά εργασίας. Και μάλιστα όχι να έχουν απλώς μια επαφή μισή ώρα στη διάρκεια μιας συνέντευξης, αλλά ε, να την... Ε, να έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή επί σειρά ημερών ε, με τους, μελλοντικ... με τους επιχειρηματίες ε, οποίους μελλοντικά ίσως ε, θα δουλέψουν έτσι ώστε να μπορέσουν να μπουν ίσως σε κάποια προγράμματα ή σε κάποιο έρασμους ή εναλλακτικά να αρχίσουν να δουλεύουν πραγματικά. Πάντως ξεκινάει με τον τρόπο αυτό μια διασυνοριακή αν θέλετε. Επαφή με άλλες χώρες και άλλες επιχειρήσεις. Δεύτερη εμπειρία της ε, του Ιδίου Πανεπιστημίου Νεότητας είναι ένα πρόγραμμα ε, σύνδεσης ε, ομάδων και οργανώσεων νέων μέσα από τα πανεπιστήμια με ομάδες βιομηχάνων και επιχειρήσεων. Βεβαίω αυτά σας τα λέω επιγραμματικά, ε, μπορώ να σας φέρω και επιπλέον στοιχεία, αλλά και αυτό το δεύτερο, αυτή η δεύτερη εμπειρία που φέρνει επαφή ανθρώπου από τι δύο ε, πλευρές ε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι τέτοιου είδου εμπειρίες μπορούν να περιληφθούν και να αποτελέσουν οδηγό και για μα Ευχαριστώ πολύ. Μπόρις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντω έκανατε μια πολύ καλή σύνοψη των πραγμάτων. Εγώ είχα την ε, ευκαιρία να βρεθώ ε, υπεύθυνο ενό προγράμματο σε μια περιφέρεια τριών εκατομμυρίων κατοίκων με ένα πρόγραμμα πάνω από με 500 φοιτητέ. Ε, εκεί λοιπόν υπήρξε σημαντική δουλειά για, την, για τον διάλογο μεταξύ ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου. Θέλουμε μια κινούμενη κοινωνία δεν θέλουμε να χάσουμε το παιχνίδι με τις ε, ε, που είναι όμως τα βασικά προβλήματα όταν μιλούμε για την ε, διαχείριση της, των επιστημών, γιατί τα αποτελέσματα της έρευνας δεν φτάνουν στις μεγάλες, δεν φτάνουν στις εταιρείε ή φτάνουν στις μεγάλες αλλά όχι στις μικρές. Ποια είναι λοιπόν τα εμπόδια που πρέπει να υπερπηδήσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το ψηλό ε, γνωστικό δυναμικό που έχουν τα, τα πανεπιστήμια. Ε, έρευνα, ας πούμε, κέντρα ερευνητικά θα μπορούσε να είναι μια λύση. Επίσης, ανταλλαγή, ανταλλαγή συνεργατών. Τα πανεπιστήμια μπορούν να διαθέτουν ε, υλικό, προσωπικό στις επιχειρήσεις και το αντίστροφο. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει και όσους είναι ιδιαίτερο ενεργοί να έχουν τις σωστές επαφές. Είναι, είναι πολύ σημαντικό νομίζω αυτό. Περίπου 90% των, επιχειρή... των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι στις, ε, στα περισσότερα ε, πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποστηρίζεται ένα ίδιο φόρουμ των οικονομικών ε, δυνατοτήτων των πανεπιστημίων. Νομίζω λοιπόν ότι ε, θα πρέπει να ζητήσουμε περισσότερα από τον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτό είναι σημαντικό και αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στην έκθεση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω ότι θα κατανοήσετε καλύτερα, θα ερμηνεύσετε καλύτερα αυτά που θα πω αυτή τη φορά, γιατί την προηγούμενη φορά δεν με καταλάβατε καλά, γιατί συμφωνούσα μαζί σας στην ουσία. Εν πάση περιπτώσει, ε, εγώ δεν θα συμφωνήσω πολύ με αυτά που άκουσα και όχι με όλα τουλάχιστον. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι το Πανεπιστήμιο εξακολουθεί να καταρτίζει νέους πτυχιούχους οι οποίοι βρίσκουν τελικά δουλειά στις επιχειρήσεις και στον επιχειρηματικό κόσμο. Οι νέοι πτυχιούχοι είναι αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν καλύτερα το θέμα της εργασίας. Δηλαδή λιγότερη ανεργία όσο ανεβαίνουμε στο επίπεδο σπουδών. Εξεπλάγει από το γεγονός ότι πολλοί συνάδελφοι αναφέρονται μονάχα στη χώρα τους και ίσως ε, πρέπει να έχουμε περισσότερη ανταλλαγή όσον αφορά τις εμπειρίες μας. Είμαι νέα βουλευτήνα και θα μιλήσω για τη χώρα μου λοιπόν. Νομίζω λοιπόν ότι στη Γαλλία το Πανεπιστήμιο έκανε, κατέβαλε εξαιρετικά μεγάλες προσπάθειες όσον αφορά τον διάλογο πανεπιστημίου επιχειρηματικού κόσμου. Και μάλιστα ε, ορισμένοι αναρωτιούνται πλέον ποια, ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του Πανεπιστημίου, σε τι χρησιμεύει το Πανεπιστήμιο. Υπάρχει ένα σημείο επί του οποίου συμφωνώ, δηλαδή τον ρόλο που πρέπει να έχουν τα πανεπιστήμια στη διαβίου κατάρτιση. Γιατί προχωράμε, ζούμε σε ένα κόσμο, οδεύουμε προς ένα κόσμο με μεγάλη κινητικότητα, νέες ανάγκες εργασίας και επομένως όσο καλύτερη και ευρύτερη γνώση έχουμε, τόσο καλύτερη δυνατότητα προσαρμογής έχουμε στις νέες συνθήκες εργασίας. Και επομένως αυτό θα πρέπει να το αναλάβει το Πανεπιστήμιο, γιατί είναι αυτό που είναι καλύτερα προετοιμασμένο έτσι ώστε να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα γιατί ε, όσο πιο εξειδικευμένη γνώση έχουμε, τόσο λιγότερη προσαρμοστικότητα έχουμε στην αγορά εργασίας. Τελευταίο στοιχείο. Διαβάζοντας ε, τον ευρωπαϊκό τύπο, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην Ευρώπη. Δημιουργούνται κινήματα στην Ευρώπη ολόκληρη σχετικά με τις ε, προτάσεις νομοθεσίες, ευρωπαϊκής νομοθεσίας όσον αφορά ε, τα θέματα που μας απασχολούν. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ε, να ακούμε τα κινήματα αυτά. Ε, μία από τις πρώτες παρεμβάσεις που έκανα ήταν η εναρμόνιση των διπλωμάτων, ήταν η δυνατότητα κινητικότητας των νέων και πιστεύω ότι εάν δεν δώσουμε σημασία στο σκέλος αυτό, τότε θα δημιουργήσουμε νέες αδυναμίες αδυναμίες κατανόηση από πλευρά των πολιτών και επομένως νέε αντιδράσεις όσον αφορά το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και τα ευρωπαϊκά σχέδια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ είμαι από το Άχεν με ένα μεγάλο πανεπιστήμιο όπου αυτά τα θέματα πραγματικά έχουν εντατικοποιηθεί σε ό,τι αφορά τη συζήτησή του. Η συζήτηση, α πούμε, για την συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τελευταίω υπάρχουν, ε, ειδικά, υπάρχουν προγράμματα συνεργασίας εταιριών και πανεπιστημίων, υπάρχουν ερευνητικά ιδρύματα, υπάρχουν συμβάσεις ερευνητικές, υπάρχουν ιδιωτικά ε, ερευνητικά ιδρύματα τα οποία συνεργάζονται με τα πανεπιστήμια. Γίνονται πολλά λοιπόν. Ένα μεγάλο πρόβλημα όμως που βλέπω είναι πέρα από τα εκτός των τεχνικών επαγγελμάτων και των τεχνικών ε, σπουδών η συνεργασία όπως είπατε το θέμα της επιχειρηματικότητας είναι πολύ δύσκολο να βρούμε ε, συνεργάτες από τον επιχειρηματικό κόσμο. Ε, ας πούμε υπάρχει μια συνεργασία σε ό,τι αφορά την ε, τελωνιακή συνεργασία. Υπάρχουν κάποια άτομα που δουλεύουν σε κάποιες, σε κάποιες επιχειρήσεις και παράλληλα σπουδάζουν. Αυτό είναι πάρα πολύ κουραστικό για του ίδιου του ε, φοιτητέ, αλλά παρόλα αυτά του δίνει τη δυνατότητα μετά να έχουν περισσότερε πιθανότητε να μπουν σε μια δουλειά. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ε, ένα διαχωρισμό μεταξύ τη βασική έρευνα και των υπολείπων επιστημών, όπου μιλούμε για ανεξαρτησία από τι επιχειρήσει και περαιτέρω εξέλιξη ανεξάρτητα από τον επιχειρηματικό κόσμο και προώθηση απλώ τη ε, βασική έρευνα. Χωρί όμω άμεση σύνδεση αυτή με την χρησιμότητά τη για τι επιχειρήσει. Η δικτύωση επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική με τις επιχειρήσεις, αλλά και η δικτύωση ε, με, τους, ε, με το κατά πόσο μπορούν οι πτυχιούχοι να μπουν σε μια καλή δουλειά. Και εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί μοντέλα τα οποία όντω λειτουργούν πολύ καλά. Α πούμε, εμεί κάνουμε ε, bonding lessons, δηλαδή ανταλλαγή εμπειριών με τι εταιρείε. Οι εταιρείε παρουσιάζονται, οι φοιτητέ έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν, να συζητήσουν με κάποιου ανθρώπου. Έτσι, σαν μια πρώτη επαφή, α πούμε. κατά διάρκεια επίση όλων των σπουδών του υπάρχει συνεργασία. Υπάρχουν υποτροφίε. Το θέμα των υποτροφιών πρέπει να βελτιωθεί στην Ευρώπη. Αν θέλουμε να, αν δούμε πραγματικά το πόσο δυναμικό υπάρχει στον τομέα αυτό, είναι μένει αχρησιμοποιητό. πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα καινούργια να, να μπορούν να τα διδαχθούν οι φοιτητέ και θα πρέπει αυτό να γίνεται στα πλαίσια των, των σπουδών του. Θα πρέπει λοιπόν αυτά, για να γίνουν όλα αυτά να του βοηθήσουμε με α, ε, ε, υποτροφίε. Επίση, τα ερευνητικά προγράμματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα ερευνητικά προγράμματα πλαίσια. και εκεί μιλούμε για την, για την συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Νομίζω λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο, πολύ σημαντικό δρόμο και το σημαντικό είναι επίση η εναρμόνιση των, κύκλων σπουδών. Δεν, είναι, δεν υπάρχει παντού αυτό. αυτό. Αν δηλαδή ένας φοιτητή πάει ας πούμε, για ένα εξάμεινο σε κάποια άλλη χώρα, πρέπει να δούμε τι γίνεται και με την αμοιβαία αναγνώριση ε, για να μην δημιουργούνται προβλήματα μετά, να μην δημιουργούνται εμπόδια. Γιατί αυτά πραγματικά δυσκολεύουν πολύ τη ζωή των φοιτητών και θα πρέπει να τους βοηθήσουμε γιατί είναι προ όφελό τους να μπορούν να συμμετέχουν σε όλα αυτά τα προγράμματα. Η εφαρμογή λοιπόν αυτή τη ε, δυνατότητα ε, σύγκριση ε, των κύκλων σπουδών νομίζω ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν καλύτερα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Σμιτ. Merci, Madame la Présidente. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Σμιτ, ο οποίος έθεσε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία προς ε, σκέψη. Ε, άκουσα να γίνεται λόγος για κοινή γλώσσα και αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έχουμε κοινή γλώσσα έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει πραγματική συνεργασία ανάμεσα στα πανεπιστήμια και τον επιχειρηματικό κόσμο. Γιατί εάν δεν υπάρχει κοινή βούληση και κοινή ε, κουλτούρα δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία. το πανεπιστήμιο και επομένως και οι διδάσκοντες θα πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Ε, θα πρέπει επομένω πρώτα να ευαισθητοποιήσουμε από τη μία πλευρά τους ε, ε, καθηγητάς και από την άλλη μεριά τους επιχειρηματίες. Βεβαίως το Πανεπιστήμιο είναι εκεί για να δίνει γνώσεις, αλλά αυτό δεν αντιτίθεται στην γνώση του κόσμου της οικονομίας. Είπατε να υπάρξουν διεύλοι επικοινωνίας, γέφυρες ανάμεσα στους δύο κόσμους και ακριβώς ακόμα και το ότι χρησιμοποιούμε την έννοια των δύο κόσμων ε, ε, σημαίνει ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα, είναι δύο διαφορετικές οντότητες τις οποίες θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε και να τους γνωρίσουμε μεταξύ μας. Ο ένας κόσμος θα πρέπει να πάει προς συνάντηση του άλλου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχω γραφεί κι εγώ στον κατάλογο. Χαίρομαι πάρα πολύ που η έκθεση αυτή παίρνει σάρκα και ωστά επιτέλους διότι πιστεύω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαζόμαστε πολύ περισσότερο. Πανεπιστήμια και οικονομία, σε όλες τις εκδοχές που αυτό μπορεί να προσλάβει. Και αυτό μπορεί να διαμορφωθεί με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Όπως επανειλημμένα ακούσαμε, μπορεί αυτό να γίνει... Ε, να υπάρχουν ε, πρακτικά ε, μαθήματα, ασκήσεις, τεχνικές τεχνολογίες... στα πανεπιστημία ή κάποιοι τομείς ε, των επιχειρήσεων να δίνουν υποτροφίες για διδακτορικά. Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν κάποιες έδρες γιατί θεωρεί κάποια επιχείρηση ότι πρέπει να χρηματοδοτήσει μία έδρα. Δηλαδή, αν χρηματοδοτεί η Mercedes μία έδρα, δεν σημαίνει ότι θα μιλάνε μόνο για τη Mercedes την έδρα αυτή στο Πανεπιστήμιο, αλλά για ένα αντικείμενο το οποίο ενδιαφέρει τους φοιτητέ και τους βοηθάει να διαμορφώσουν το μέλλον τους και να το προσανατολίσουν αλλιώς πολλοί φοιτητέ γνωρίζουν πάρα πολύ λίγα, πολύ λίγα ελάχιστα για την οικονομία, για το τι θα μπορούσαν να κάνουν στο μέλλον. Στο πανεπιστήμιο συχνά δεν τους ε, προσανατολίζουν, δεν τους βοηθάνε, δεν υπάρχει πρόταση ε, ε, για κάτι το διαφορετικό από αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα. Μπορεί λοιπόν να υπάρχει μια ανταλλαγή. Το κάνουμε αυτό με τον έρασμο και το πήραμε από το Λεωνάρδο αυτό, ε, με τις ε, ασκήσεις, ε, τις περιόδους άσκησης δηλαδή στις επιχειρήσεις. Υπάρχει ήδη στον έρασμα αυτό. Αλλά μήπως να σκεφτούμε οι επιχειρήσεις, οι μάνατζερ να πηγαίνουν και ως επισκέπτες καθηγητές στα πανεπιστήμια και να διδάσκουν ή να παρουσιάζουν την κατάσταση που ζουν ήδη στην πράξη. Και ε, κάποιος φοιτητής μπορεί να πάρει μια ιδέα ότι α, αυτό μου κάνει, για να το κοιτάξω και αυτό. Να ανοίξει αυτό το πανεπιστήμιο, να μην είναι ένας πύργος φιλτισένιος. Ε, αυτό έχει γίνει σε πολλούς τομείς. Να σας πω από το δικό μου τομέα που το ξέρω, ε, όχι για να περιευθολογήσω, αλλά να θυμίσω ότι το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου έχει στηθεί ολόκληρο ε, με βάση αυτή την ιδέα ή το Campus Europe, αυτή η συνεργασία των πανεπιστημίων μεταξύ ε, των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Υπάρχουν πολλά θαυμαστά ε, παραδείγματα και χαίρομαι που αναφέρετε και εσείς παραδείγματα από τα κράτη σας, διότι ακριβώς με τις βάλτιστες πρακτικές και μόνο θα έχουμε καλά ε, πορίσματα και αποτελέσματα. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει παντού σε ίδιο επίπεδο ή ταυτόχρονα. Αλλά στην έκθεση να πούμε ποιες είναι οι δυνατότητες που υπάρχουν για να εμπλουτίζουμε. Η κυρία Βερζιά μίλησε για τους φοιτητέ και βεβαίως να ακούμε και τους φοιτητέ. Αλλά οι φοιτητέ, ας πούμε, στη Γερμανία που βγαίνουν τώρα στους δρόμους, γιατί βγαίνουν στους δρόμους κυρίως, διότι ε, να βάγισε το σχέδιο της Μπολόνια. Και πριν από ένα μισή χρόνο εγώ είχα κάνει εδώ στην έκθεση ε, για την Πολόνια, παρόλο που δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι, ε, τα κράτη-μέλη και Κάποιοι άλλοι θέλησαν να κάνουν την Πολόνια ρήμη του κοινοβουλίου. Αν το είχαν περάσει από το κοινοβούλιο θα είχαν αποφύγει ε, αυτές τις παιδικές ασθένειες. Και βγαίνουν φοιτητέ στους δρόμους ε, γιατί δεν μπορούν να κυκλοφορούν, να έχουν την κινητικότητα. Όταν ε, μου συμπυκνώνει ένα πτυχίο πενταετέ σε τρία χρόνια, πού να προλάβω να πάω και στο εξωτερικό να κάνω κανένα εξάμεινο. Και έχουν δίκιο φοιτητέ και βγαίνουν στους δρόμους. Να πω και ένα άλλο παράδειγμα. Στο Βερολίνο έχουμε δύο μεγάλα πανεπιστήμια, το Humboldt και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο. Στο παρελθόν μπορούσε ο καθένας να σπουδάζει, να πάρει διάφορες θεματικές ενότητες από το ένα πανεπιστήμιο και το άλλο. Για να κάνεις τον Μπάτσελο λοιπόν της Μπολόνια σήμερα, αν είσαι γραμμένο στο Humboldt, μόνο στο Humboldt, στο ελεύθερο όχι. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτή η πλήση ε, η, σχολική προσέγγιση του πανεπιστημίου. Τι θέλησαμε αυτό το μπάτσελορ της Μπολόνια, το πτυχίο. Ε, ε, αυτό που θέλησαμε δεν το πετύχαμε. Και για τη συνεργασία και πάλι των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να δούμε και το bachelor, το πτυχίο και το master, το μεταπτυχιακό, να το εξετάσουμε καλύτερα και να ακούμε για τους φοιτητέ που μας τα λένε κάθε μέρα γιατί ε, υποφέρουν από αυτή την κατάσταση τα δίνα. Λοιπόν, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Παλ Σμιτ, θα ήθελα να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Μπερνάντο Ντεκουερός, να μας πει την άποψή της. Παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή σύνοψη του περιεχομένου της ανακοίνωσης της Επιτροπής. Όπως ορθώς είπε ο εισηγητής στην αρχή της ομιλίας του, η στήριξη των κρατών μελών ε, ως προς τον εξυγχρονισμό των πανεπιστημίων είναι ένας από τους πυλώνες, από τα κυρίαρχα στοιχεία της ε, Λισαβόνας γιατί θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε μια κοινωνία η οποία θα βασίζεται στη γνώμη. Τώρα, ακρογωνιαίος λήθος ε, της όλης προσέγγισης αποτελεί και η διασύνδεση ανάμεσα στα πανεπιστήμια και τον επιχειρηματικό κόσμο. Το είπατε άλλωστε κι εσείς ε, ότι τα πανεπιστήμια θα πρέπει να ανοίξουν περισσότερο προς τις, και να, για να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες ε, της ε, κοινωνίας και επομένως έχουν δημιουργηθεί και εργαλεία όπως το Φόρουμ Πανεπιστημίων Επιχειρηματικών επιχειρήσεων και με την ανακοίνωση της Επιτροπής προσπαθεί να απαντήσει σαφέστερα. Τα πανεπιστήμια είναι σημαντικός πόλος γνώσης, έχουν σημαντική δυνατότητα ε, πρόθεσης της έρευνας και της καινοτομίας, αλλά ξέρουμε ότι το δυναμικό τους δεν το χρησιμοποιούμε 100%. Στο, στην ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρεται ε, σε έξι ε, στοιχεία. Νέα, ε, νέο πρόγραμμα σπουδών, νέα διακυβέρνηση, διασύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο. Επίσης θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι αλλαγές στην αγορά εργασίας θα πρέπει να αλλάζουν και το πανεπιστήμιο και το περιεχόμενο σπουδών τους. Δεν είναι δυνατόν πτυχιούχοι να βγαίνουν χωρίς να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες ε, της, ε, ε, του επιχειρηματικού κόσμου και επομένως τα πανεπιστημιακά προγράμματα θα πρέπει να οικοδομηθούν με τρόπο τέτοιο ώστε να δίνουν τη δυνατότητα στους πτυχιούχους να μορφώνονται σίγουρα αλλά και να βρουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Οι επιχειρηματίες από την άλλη πλευρά έχουν την υποχρέωση ε, να ε, ε, δημιουργούν τις προϋποθέσεις αυτές έτσι ώστε οι πτυχιούχοι να μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που που ευθύνεται για την ε, ε, κακή κατάσταση όσον αφορά τη διασύνδεση επιχειρηματικού κόσμου και πανεπιστημίου είναι η μειωμένη επιχειρηματικότητα ε, στην Ευρώπη. Σε γενικές γραμμές βλέπουμε ότι είναι μικρότερη η βούληση για επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη. Επομένως, θα πρέπει να ανταποκριθούμε στην πρόκληση η οποία θέλει να αναπτυχθεί αυτή η επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη. Βεβαίως θέλουμε σπουδαστές οι πτυχιούχους που θα έχουν γνώσεις ε, και οι οποίοι θα είναι εύκολοι όσον αφορά την κινητικότητα και ε, που θα έχουν την ε, επιθυμία να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει οι πτυχιούχοι να κατανοούν τις εξελίξεις στον, στην αγορά εργασίας και στον επιχειρηματικό κόσμο. Βεβαίως η μεταφορά γνώσης ε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Καλύτερη επαφή, αμοιβαία αναγνώριση ε, διπλωμάτων, αμοιβαία αναγνώριση ακαδημαϊκών περιεχομένων που θα μπορέσουν να δώσουν ε, έναυσμα πραγματικό σε μια νέα, σε μια ανάπτυξη καλύτερη που θα βασίζεται στη διαβίου κατάρτιση. Η επιχειρηματίες, ή επιχειρήσεις από την άλλη πλευρά θα πρέπει να απομονώσουν τις ανάγκες τους ε, και ε, να μεταφέρουν λοιπόν τις ανάγκες αυτές ή στα πανεπιστήμια. Η τα πανεπιστημια η δημιουργια των business forums υπογραμμίζουν την επιθυμία θεσμοθέτησης ε, σχέσεων και βεβαίως αυτές οι σχέσεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση καλής συνεργασίας ανάμεσα στα πανεπιστήμια και τον επιχειρηματικό κόσμο καλή συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους, σε όλους τους εμπλεκόμενους, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ε, ε, πληθώρα δυνατοτήτων ε, στις οποίες θα βασιστούν οι νέες σχέσεις και οι νέες συνεργασίες. Συνεργασίες οι οποίες θα παρουσιάζουν οπωσδήποτε μεγάλη προστιθέμενη αξία και για τα πανεπιστήμια και για τους καθηγητές και για τους φοιτητές αλλά κατ' επέκταση και για τον επιχειρηματικό κόσμο και για την κοινωνία το να φέρουμε κοντύτερα ε, την, τον επιχειρηματικό κόσμο, τον κόσμο της εργασίας με τον κόσμο των σπουδών, ε, μας δείχνει το δρόμο καλή εταιρική συνεργασία, καλή συνεργασία, συνεργασία σε εταιρική σχέση. Θα δώσει τη δυνατότητα ε, και σε δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες και στις δημόσιες αρχές και στην κοινωνία και στους πολίτες ε, ε, εν γέννη, είτε είναι καθηγητές, είτε είναι φοιτητές, είτε είναι επιχειρηματίες, θα δώσει καλό αποτέλεσμα σε όλους. Είναι μια κατάσταση win-win. Θα πρέπει βεβαίως να καλύψουμε και όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και όλους τους στο τομείς του επιχειρηματικού κόσμου, να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκά εργαλεία τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να υλοποιηθούν ε, οι αρχές αυτές. Τα επόμενα ε, φόρα είναι τα εξής θεματικό φόρουμ ε, συνεργασίας με το ETF, φόρουμ στην Τσεχική Δημοκρατία τον Φεβρουάριο διεύρυνση του φόρουμ σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο και ένα τελευταίο φόρουμ τον Μάιο του 2010. Πιστεύουμε ότι η εργασία των ε, φόρα ε, αυτών που ανέφερα μπορούν να δημιουργήσουν κινητικότητα ε, και να κινητοποιήσουν επομένως δράσεις σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, ε, κύριε Σμιτ. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ακριβώς ε, αυτό που περίμενα συνέβη. Πολύ χρήσιμα σχόλια, πολύ χρήσιμες προτάσεις και αμέσως ε, καταλαβαίνει κανείς ότι το θέμα αυτό κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση σε όλα τα κράτη-μέλη, διότι η ζήτηση και η προσφορά δεν συναντιόνται. Γι' αυτό έχουμε τόσους άνεργους πτυχιούχους με τόσο υψηλή ενεργεία. Δεν θυμάμαι ποιος το είπε, ε, αλλά κάποιος ανέφερε ότι τα πανεπιστήμια αναλαμβάνουν τεράστια ευθύνη για τους πτυχιούχους τους που παράγουν. Τι τους κάνουν, τους δίνουν την τίβενο, τους φοράνε και ένα καπέλο, τους φύγουν και το χέρι συγχαρητήρια από φοιτής, δεν χαίρεται. Και από εκεί και πέρα δεν ενδιαφέρεται το πανεπιστήμιο να μάθουν τι απογίνονται αυτοί οι άνθρωποι. Βρίσκουν δουλειά, τι κάνουν στη ζωή τους. Ευχαριστώ λοιπόν ε, τους συναδέλφους, δεν θέλω να πω στις λεπτομέρειες των όσων αναφέρεται, ε, καλές πρακτικές, καλά παραδείγματα, βέλτιστες πρακτικές τις λέμε, δεν ξέρω αν ε, χωρούν ε, όλα αυτά σε μία έκθεση, αν μπορώ να μπω σε τόσες λεπτομέρειες, θα το συζητήσουμε αργότερα. Ε, από τη δημόσια ακρόαση δεν περισσότερα περιμένω από ότι από την έκθεση. Θα έχουμε εκεί πριτάνεις, καθηγητές πανεπιστημίου, διδακτικό προσωπικό, ακριβώ αυτές οι βέλτισες πρακτικές να μας ενημερώσουν τι συμβαίνει. Συμφωνώ και με τον κύριο Λάκεγκαρτ που λέει ότι τα Υπουργεία Παιδείας θα πρέπει να συνεργάζονται με τα ε, Υπουργεία Απασχόλησης και να συμμετέχουν στη διαβούλευση. Επίσης, ένα πολύ καλό εργαλείο θα ήταν οι υποτροφίες ενδεχομένω. Συμφωνώ ότι στη διαδικασία αυτή δεν μετέχουν πολλοί φυσικές επιστήμες, ε, δεν ενδιαφέρονται πάρα πολύ ε, για τη συνεργασία με την οικονομία, αλλά οι φυσικές επιστήμες είναι εξίσου σημαντικές όπως είναι και ε, οι τεχνολογίες, η μηχανική, τα πολυτεχνία, η κοινωνία της προφορίας κτλ. Το γεγονός τώρα ότι θα μπορούσαν τα πανεπιστήμια να συνάπτουν και συμβάσεις με τους φοιτητές. Πολύ καλή ιδέα και συμβάλλει πολύ και στην αυτοπεποίθηση των φοιτητών. Από εκεί και πέρα ακούσαμε και κάτι για την ποιότητα των πανεπιστημίων. Θα πρέπει να είναι δυναμικά, να συμβαδίζουμε τις αλλαγές που παρατηρούμε και στον επιχειρηματικό κόσμο. Δηλαδή θα πρέπει να είναι σε θέση και τα πανεπιστήμια να νεώνονται και να ε, ξεχρονίζονται. Και συμφωνώ με την εγκάρση λεγόμενη χρηματοδότηση, δηλαδή ε, να πάρουμε ε, ε, ιδέες και συμμετοχή ε, εργαζομένων στις επιχειρήσεις στα πανεπιστημία που να δίνουν διαλέξεις, αλλά και το αντίστροφο, καθηγητές στις επιχειρήσεις. Επίσης ακούσαμε για περίοδους άσκησης σε επιχειρήσεις και τελειώνω πρόεδρε με το εξής που θέλω να σας πω. Επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα Ζούσα σε μια σοσιαλιστική χώρα που είχαμε πολλές ελλείψεις και είχα μπει σε ένα κρεοπολείο που δεν είχε πάντα πολύ κρέας και εγώ χαιρετούσα πάντα ε, εγκάρδια τον κρεοπόλιο, εκείνος δεν ήταν χαρούμενος. Ε, γιατί είχε πολλούς πελάτες αλλά δεν είχε κρέας. Τώρα που πάω στο κρεοπολείο, χαρά να δείτε που κάνει ο κρεοπόλης. Κύριε Σμιτ, καλωσορίσατε. Γιατί τώρα τι έχουμε, έχουμε μεγαλύτερη ζήτηση και λιγότερη προσφορά. Ε, συγγνώμη, μεγαλύτερη προσφορά και λιγότερη ζήτηση. Στο παρελθόν που χαιρόμουν εγώ που τον έβλεπα και εκείνο